Right, welcome everybody. Καλώς ήλθατε όλοι. Βλέπω ότι μάλλον κάποιοι συνεχίζουν το χριστουγεννιάτικο τους ε, γεύμα ή κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, σας ζητώ να εγκρίνετε την ημερησία διάταξη, δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Αν εφαντήρησαν εγκρίνεται λοιπόν. Έχουμε πολλές ανακοινώσεις από την Πρόεδρο. Καταρχήν είμαστε στο διαδίκτυο, το ξέρετε αυτό. Δεύτερον, όπως είπε ήδη η γραμματεία σε εσά. η συνεδρίασή μας αύριο την Τρίτη θα είναι στο aasp 3 Ή δύο τι ειπε Και σας ε, θυμίζω λοιπόν, στο τέλος της συνεδρίασης να πάρετε τους φακέλους σας, γιατί δεν θα είμαστε εδώ αύριο. θα γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας με την Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων. Στις 20 Δεκεμβρίου, αύριο δηλαδή, 6.30 με 8, δηλαδή μετά από το τέλος της συνεδρίασής μας, δεν είχαμε άλλο σλότ για μια κίνηση συνεδρία των δύο επιτροπών. Αυτά είναι τώρα ανακοινώσει του Πρόεδρου Ζωαμπόλ. να πεις κάτι παρόλα αυτά μια διευκρίνηση. Δεν είναι στις 10 όπως γράφει η γραμματεία, είναι από τις 6.30 ως τις 8 η κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, έτσι δεν είναι. 6 και 30 με 8 λέει η πρόεδρος. 6.30 με 8 λοιπόν. Μόλις τελειώσουμε την ε, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά, αν θέλει ο Χιαραμπής, θα τελειώσουμε στις 8 η ώρα την κοινή συνεδρίαση. Στο 6Q2 γίνεται αυτό, η κοινή συνεδρίαση. Άλλη αίθουσα από αυτή όπου θα συνεδριάζουμε. Θα πρέπει να τρέξουμε από το SP3G2 ε, στο 6Q2 που απέχει παρασάγκας για να μπορέσουμε να είμαστε στην κοινή συνεδρίαση. Δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να έχουμε διακτηνισμό, αλλά θα τα καταφέρουμε. Πού θα πάει έχει διανεμηθεί ήδη ένα σχέδιο του σχεδίου συνθήκης, ένα αντίγραφο του σχεδίου συνθήκης σε όλους. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε, θα γίνει φυσικά μετάδοση στο διαδίκτυο όπως είναι φυσιολογικό. Στις 12 Δεκεμβρίου πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συζητήσαμε τον κύριο Ντράγκη και το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα ανοιχτό και εγκάρδιο κλίμα για τον ο ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας στην κρίση κρατικού χρέους και για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε 9 Σεπτεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συζητήσαμε, εστιάσαμε περισσότερο στα θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και φυσικά ο Μάριο Ντράγκη θα έρθει αργότερα σήμερα. Και αύριο το πρωί θα κάνω κάποιες ανακοινώσεις για διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 73 εφόσον η Κορεπέρ μας επιβεβαιώσει ότι θα στείλουμε πράγματι αυτό το κείμενο και μετά για τον τρίλογο για τα παράγωγα. Ο προηγούμενος τρίλογος έγινε στις 12 Δεκεμβρίου ήταν ο τέταρτος, ο πέμπτος έλαβε χώρα σήμερα το πρωί. Υπήρξε πρόοδος, έχουν μείνει μερικά εκκρεμή θέματα και ελπίζουμε ότι στις 23 Ιανουαρίου θα γίνει ο επόμενος τριγωνικός διάλογος. Κάποια στιγμή αργά το απόγευμα, νωρίς το, αργά το πρωί, νωρίς το απόγευμα, πρώτο σας αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Περνάμε τώρα στο θέμα 3 που είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών καθώς και Περιφερειακών Λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η συγγήτρια είναι η κυρία Σάρον Μπάουλς, εξ της Επιτροπής μας. Το σχέδιο έκθεσης έχει διανεμηθεί, όπως είπα, στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, την προηγούμενη φορά πριν από ένα μήνα. Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει τους κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούνται για τη συμπίληση και την δημοσίευση το λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρόταση της Κομισιόν ουσιαστικά σημαίνει μια σημαντική μεταρρύθμιση του συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας την τροποποίηση του συστήματος του ΟΗΕ για τους εθνικούς λογαριασμούς γνωστού ως SMA, που ενεκρίθη το 2008. Προσπάθησα να καλύψω μια σειρά από σημεία σε αυτή την έκθεση. Καταρχήν ότι τα κράτη-μέλη έχουν ε, εκφράσει ανησυχίε για το διοικητικό άχθος και το προβάλλουν αυτό ως αίτιο εξαιρέσεων και ένα από τα πράγματα τα οποία έπραξα είναι να προτείνω ότι για το μέλλον θα πρέπει να βρούνε αυτόματους και ε, πραγματικού χρόνου μηχανισμούς συλλογής στοιχείων ώστε να μπορούν τα στατιστικά στοιχεία να έρχονται άμεσα από παραγωγικά τα ταμεία των ε, σούπερ μάρκετ. Και ένα άλλο σημείο το οποίο τόνισα είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο πλήρη για να έχουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, Ιδίω σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς του δημόσιου τομέα και θα πρέπει να δημοσιεύονται έχοντας υπόψη τον τελικό χρήστη. Επίσης υπογράμμισα ότι χρειάζεται περαιτέρω μεθοδολογική εργασία για να καταλήξουμε σε μια πληρέστερη απεικόνιση των περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων των οικοκυριών και του δημόσιου τομέα. Ξέρω ότι αυτό ενδιαφέρει κάποιο σκιώδη εισηγητή. Προσπάθησα να μειώσω τι εξαιρέσει στο απολύτω απαραίτητο και επίση να θέσω χρονικά όρια στη διάρκεια αυτών των εξαιρέσεων. Ένα λόγο εξαιρέσεων στο παρελθόν ήταν η ανεπάρκεια πόρων, αλλά ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να μείνει σε μια τέτοια κατάσταση στο δίνεκες, θα πρέπει να βρει μια λύση για τα θέματα αυτά. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτή η δικαιολογία δεν μπορεί να μείνει ανοιχτή για πάντα. Επίσης ζητούμε από την Κομισιόν να ε, διατυπώσει το πρόγραμμα για την ε, διαβίβαση δεδομένων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο σε αυτό το πρόγραμμα και δεν κατανοούν απόλυτα τα κράτη-μέλη ποιε είναι οι υποχρεώσει του σε σχέση ιδίω με τι καταληκτικέ προθεσμίε για τα στατιστικά στοιχεία. Αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθεί επίση το Συμβούλιο. να υπάρχει και έκθεση ποιότητα από την Κομισιόν προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για του Εθνικού Λογαριασμού κάθε δύο χρόνια και επιτρέπει, όπω ε, πάντα έχουμε κάνει, να υπάρχει και ένα μεγαλύτερο χρόνο εξέταση για τι κατά ε, εκχώρηση πράξη τρει μήνε αντί για δύο. Και άλλαξα το λεγόμενο κριτήριο του 50% για τους λογαριασμούς του δημόσιου τομέα, ώστε τώρα να λέγεται κριτήριο του 100%. Με το κριτήριο του 50%, τον κανόνα αυτό, οι εταιρείε οι οποίες έχουν κρατική συμμετοχή είτε τοπικού είτε κεντρικού επίπεδου, καταγράφονται στον κεντρικό τομέα μόνο εάν οι πωλήσει τους δεν καλύπτουν τουλάχιστον το ίμιση του κόστους της λειτουργίας τους. Παραδείγματος χάρη μια υπηρεσία τοπικών μεταφορών, αν παίρνει 51% των ε, εξόδων της από πωλήσει, τότε θεωρείται ότι είναι εταιρεία ιδιωτικού τομέα. Αυτό όμως δεν αντανακλά πραγματικά την κατάσταση. Μια εταιρεία η οποία δεν μπορεί να καλύψει τα 100% του κόστους παραγωγής της με τα έσοδά της δεν λειτουργεί σαν μια εταιρεία η οποία μεγιστοποιεί το κέρδος της και επομένως δεν θα έπρεπε κατά τη δική μου άποψη να ταξινομηθεί ως ιδιωτική εταιρεία, εταιρεία ιδιωτικού τομέα. Μια λύση στο πρόβλημα αυτό θα ήταν να αλλάξουμε τη μεθοδολογία και να διευρύνουμε το, την περίμετρο της γενικής κυβέρνησης περιλαμβάνοντας δημόσιους φορείς στο δημόσιο τομέα, όλους τους φορείς λοιπόν στο δημόσιο τομέα. Γι' αυτό ζητώ να άρουμε το κριτήριο του 50% και να έχουμε το κριτήριο του 100%. Οπότε όλες συμπούρμπουλες οι εταιρείε αυτές είναι στο δημόσιο τομέα. Και καταθέτω και τροπολογίες οι οποίες έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχω ενσωματώσει όλες τις προτινόμενες τροπολογίες τους μαζί με την αιτιολόγηση που περιλαμβάνουν γιατί νομίζω ότι είναι ορθό και πρέπει να τη συζητήσουμε σε αυτό το χώρο και γενικά συμφωνώ μαζί τους και προσβλέπω να ακούσω την άποψη των σκιωδών εισηγητών για τις δικές μου τροπολογίες και αυτές που έχω συμπεριλάβει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο θέλει να λάβει το λόγο, αλλά έχουμε και κάποιους σκιώδεις ηγητές. Θεόδωρο, θες να λάβεις το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε μου. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς για τις προσπάθειές σας και να υπενθυμίσω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι πάνω από χίλιες σελίδες. Εξέτασα τις τροπολογίες σας και νομίζω ότι τις περισσότερες μπορούμε να τις δεχτούμε. Συμφωνούμε με τις αποσαφηνήσεις σας για τις εξαιρεσει που πρέπει να είναι προσωρινές και να αναθεωρούνται τακτικά. όσο για την έκθεση που υπέβαλε η Κομισιόν στο Κοινοβούλιο για την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων από τους εθνικούς και περιφερειακούς προϋπαλογισμούς. Νομίζω ότι τέτοια έκθεση πρέπει να γίνεται κάθε τρία χρόνια, όπως γίνεται για άλλα θέματα, για τα οποία υποβάλλει η έκθεση Κομισιόν στο Κοινοβούλιο. Αυτά τα λέει η τροπολογία 11. Για το 50% του κόστους τώρα, νομίζω ότι θα επέτρεπε αυτό και σε ιδιώτες και σε κρατικές οντότητες να, να, να. Τέλεια. Πρέπει όμως να εξετάσουμε περαιτέρω το κείμενο για να δούμε γιατί προτείνει η Κομισιόν αυτό το 50%. Όταν λέει ότι κάποτε πρέπει να φτάσουμε το 100% τι εννοεί. Υπάρχουν πολλές δημόσιες υπηρεσίες που έχουν επιχορηγήσεις κρατικές όπως το νερό, η μεταφορά επιβατών, οι συγκοινωνίες κλπ. Και η τιμή που πληρώνουν οι πελάτες και πελάτησες δεν καλύπτει 100% του κόστους. Τροπολογία 19 τώρα προτείνει διαγραφή. Είναι η τροπολογία της ΕΚΤ. Το συζητήσαμε και στην ομάδα μας εμείς και νομίζουμε ότι δεν θα θέσει ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά θέλουμε να δούμε τι θα πούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι της Επιτροπής. Λοιπόν, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε λοιπόν, μέχρι τώρα, τουλάχιστον για τη δική μου χώρα, μου φαίνεται ότι τίθεται ένα θέμα προθεσμιών που αναφέρονται στην προσθήκη. Εκεί φαίνεται υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ χωρών μελών και πρέπει να γίνουν και άλλες διαβουλεύσεις. Θα πάνε αντιπροσωπείες του Eurostat να δουν στα κράτη-μέλη γιατί δεν είναι οι ίδιες οι περίοδοι που προβλέπονται για όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά επειδή όπως σας είπα είναι πολύ μακρύ κείμενο, νομίζω κυρία εισηγήτρια ότι εργαστήκατε πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Φίλιππε θέλεις να μιλήσεις. Ορίστε, ο Φίλιππος. Και μετά ο Ούγος. Α, όχι. Εγώ αντικαθιστώ την κυρία Κέι, η οποία συμφωνεί απόλυτα ότι πρέπει οι πολίτες να έχουν αξιόπιστα στοιχεία, πράγμα που δεν ίσχυε για πολλά κράτη-μέλη και συνέβαλε η ανομαλία αυτή στην τωρινή κατάσταση. Άλλο είναι να εγκρίνεται νομοθεσία και άλλο να εφαρμόζεται. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε τεράστιο πρόσθετο γραφειοκρατικό κόστος στις χώρες μέλη. Και ορισμένες γι' αυτόν τον λόγο έχουν αντιρρήσεις ότι θα λειτουργήσουν οι προτάσεις της ΕΚΤ. Και το Συμβούλιο και η ΕΚΤ πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα είναι εφαρμόσιμα αυτά που πρατείνουν ο Φίλιππος. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα θέλω να υποστηρίξω κάποιες από τις τροπολογίες που υπέβαλε Σάρων όσον αφορά τη διαφάνεια και προσβάσει στις πληροφορίε και ενδιαφέρουσε πληροφορίε που πρέπει να δίνονται στου εμπλεκομένου φορεί και στου πολίτε. Είναι πρόσδεκτο το ότι τονίζει την ανάγκη να καταγράφονται και οι δαπάνε ε, των ερευνών σαν ε, σταθερό κεφάλαιο, τι να πω, ανόητε δαπάνε, πώ να το πω, σαν τακτικέ δαπάνε, κανονικέ δαπάνε, στι τροπολογίε 3 και 6 αναφέρεσαι την ανάγκη διενέργειας περισσότερων μεθοδολογικών μελετών ούτως ώστε να δούμε τι γίνεται στον τομέα του περιβάλλοντος. Αυτό που αποκαλούμε ΑΕΠ και πέρα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Παίρνεις αυτό που υπολογίζεις και αυτό που στους υπολογισμούς. Πρέπει να αποσαφινιστεί το κείμενο σε αυτά τα σημεία. Αλλά πέραν τούτων ε, είμαστε ικανοποιημένοι με τις τροπολογίες που προτείνεις. Καλώς. Άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Ο κ. Σουκλούνα είναι σε άλλη συνεδρίαση, οπότε δεν μπορεί να είναι παρόν εδώ. Οπότε υποθέτω θα μου γνωστοποιήσει τις απόψεις του, αν δεν εμφανιστεί. Για να προχωρήσουμε, να στραφώ προς τον κύριο Νόρντλαντ, εκπρόσωπο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Νόρντλαντ, διευθυντής της ε, Eurostat. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι θα για την υποστήριξη της Επιτροπής όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Υποστήριξη όσον αφορά την ουσία, όπως αποδεικνύεται το σχέδιο εκθέσεως που μελετήσαμε, όσο και όσον αφορά και το χρονοδιάγραμμα που καταρτήσατε, διότι ταιριάζει άριστα με την ανάγκη εφαρμογής των προτύπων στα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν τρία σημεία που θέλω να αναφέρω για την ουσία της έκθεσης. Συμφωνούμε απόλυτα με την ανάγκη να περιοριστούν κάποιες παρεκκλήσεις που δίνονται στα κράτη-μέλη βάσει του κειμένου. Είναι σαφές ότι τη στιγμή που θα δώσουμε πολλές παρεκκλήσεις, αν το κάνουμε αυτό, η αξία όσον αφορά τα συγκρίσιμα στατιστικά μειώνεται άμεσα. Και γι' αυτό στην πρότασή μας έχουμε περιορίσει τις υποθέσεις όπου δεχόμαστε παρεκκλήσεις, όπου η κατάσταση πραγματική των κρατών μελών απαιτεί μεγάλη προσαρμογή των συστημάτων τους, των στατιστικών στοιχείων και θα θέλαμε εκεί να μείνουμε, να μην ανοίξουμε την πόρτα και για άλλες περιστάσεις, όπως μεθοδολογικά προβλήματα ή παρεμφερή προβλήματα. Δεν θεωρούμε ότι αυτός είναι ένας λόγος για εξαιρέσεις. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι αυτό που και εσείς και κάποιοι από τους άλλους που πήραν το λόγο έθιξαν. Δηλαδή το θέμα του διαχωρισμού δραστηριοτήτων αγοράς και δραστηριοτήτων εκτός αγοράς. Δεχόμαστε μεν την αξία του επιχειρήματος υπέρ της αλλαγής 100% είναι μάλλον ευαίσθητο ζήτημα. Σας προειδοποιώ ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν κάποιες απόψεις από αυτού στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Και το τρίτο αφορά κάποιες στοιχείες που αφορούν τα θεσμικά όργανα, θεσμικά θέματα συμπεριλαμβανομένων και των ανεπισήμων διαβουλεύσεων με την ΕΚΤ στις κατεξισοδότησης πράξεις. Ελπίζουμε το τελικό αποτέλεσμα να είναι κάτι που θα ευθυγραμμίζεται με τις διοργανικές συμφωνίες που έχουν θεσπιστεί σε πλέον οριζόντιο επίπεδο, αγαστές, άριστες οι σχέσεις μας οι καθημερινές με την ΕΚΤ, όμως θα ελπίζαμε να βρούμε λύσεις οι οποίες δεν θα απαιτούν υπερβολική γραφειοκρατία. Στόχος εξάλλου είναι η ευελιξία όσον αφορά τις εξουσιοδότησης ε, πράξης, ούτως ώστε να προσαρμόσουν αλλαγές στον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ παρόλα αυτά για αυτά που προτάθηκαν και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους σκιώδεις που μπόρεσαν να έρθουν στις προηγούμενες συναντήσεις και μπορέσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις πριν από την παρουσίαση της εκθεσής μου. Θα ήθελα και πάλι να μιλήσω για τον κανόνα του 50%-100%. Και εγώ δεν ήθελα την ιδέα του να υπάρχει μια αλλαγή στο 50%. Ήθελα να συμπεριλάβω το στοιχείο αυτό ως κομμάτι του δημοσίου τομέα. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις δηλαδή είτε καλύπτουν το 50% ή όχι. Τώρα αν μπορεί να γίνει αυτό ή όχι, αν μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του 50% αλλά να κατά κάποιο τρόπο να υπάρξει και κάποια απομείωση σε σχέση με το 100% δεν ξέρω. Όπως είπε και ο Τίοντο, υπάρχουν πολλές εταιρείες που υπάρχει κρατική συμμετοχή. Αν δεν καταγράφουμε την δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων, αυτό είναι λανθασμένο. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό για να αντιμετωπίσουμε πλήρως την πραγματικότητα. Για το κόστος κάποιων προτάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το γνωρίζω αυτό και γι' αυτό αναφέρω αυτές τις προτάσεις για βάση συζήτησης. Πρέπει όμως να τα εξετάσουμε όλα αυτά και να κάνουμε μια ανάλυση κόστους οφέλους. Νομίζω ότι θα ήταν ορθό, τουλάχιστον καταρχήν, να αναγνωρίσουμε την ανάγκη να υπάρχουν επακριβή στατιστικά στοιχεία λόγω των συνθήκων στις οποίες βρισκόμαστε και αυτό νομίζω ότι έχει την υποστήριξη της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι αν τελικά καταδειχθεί ότι κάποιες από τις αιτήσει αυτές της Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να έχουν δυσβάστακτο κόστος, θα πρέπει να τις αλλάξουμε. Αλλά και πάλι όλα αυτά τα οποία πρότεινα ήταν με διαβούλευση με την Κεντρική Τράπεζα και θα προσπαθήσω να βρω κάποια διατύπωση η οποία συνάδει με τη διαθεσμική συμφωνία γιατί πάντα για τα στατιστικά στοιχεία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι από τους κυριότερους χρήστες αυτών των στοιχείων. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να βρούμε την κατάλληλη διατύπωση η οποία μας ικανοποιεί για το σημείο αυτό. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Η προθεσμία των τροπολογιών είναι 18 Ιανουαρίου το μεσημέρι. Στις 28 θα συζητήσουμε στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε στις 20 Μαρτίου στην Επιτροπή μας και το Μάιο, αν θέλει ο Θεός, θα πάμε στην Ολομέλη. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ακολουθεί στη μέση διάταξη η έκθεση της κυρίας Αστρίδ Λούλινγκ, η οποία δεν είναι εδώ όμως. Είναι έξω. Μήπως μπορεί κάποιος να την ειδοποιήσει ότι έρχεται η ώρα της. Ναι, 10 λεπτά πιο νωρί τελειώσαμε στο σημείο αυτό το πρώτο. Ναι, ναι, Αστρίδη, συγγνώμη, απλώς ε, προτρέξαμε λιγάκι. Όλοι είναι εδώ. Ο Φελίπ. Η Εύα δεν είναι. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 4. Φορολογία ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας, αναδιάθρωση του κοινοτικού πλαισίου, του ενωσιακού καλύτερα. Εξετάζουμε τις τροπολογίες. Και η συντάκτρια, η συγγήτρια μάλλον, είναι η Αστρίδ. Μόλις τακτοποιήσει τα χαρτιά της μπορεί να ξεκινήσει. Δεν σε πιέζουμε γιατί έχουμε τελειώσει νωρίς το προηγούμενο θέμα. Μόνο 219 τροπολογίες έχουν καταθέσει τα μέλη της Επιτροπής. Υπήρξε αρκετή λοιπόν δραστηριότητα για τα θέματα αυτά. Yes, five opinion giving committees, so that... Έχουμε πέντε γνωμοδοτικές επιτροπές. Οπότε μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά. ready. Οπότε θα σας τρίδω. Μα έτοιμη, έτοιμη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και με συγχωρείτε αλλά προχωρήσατε πολύ γρήγορα μου είχατε πει παρατέταρτο τέλος πάντων έτσι θα έχουμε περισσότερο χρόνο περίμενε λίγο ο Ιωάννης Παύλος. Στο τρία δεν ακούω γαλλικά αλλά κάποια άλλη γλώσσα. <laughs> Μα είναι τα δικά μου γαλλικά που δεν τα καταλαβαίνεις. Γι' αυτό. Ιταλικά είναι κάτι τέτοιο είναι. Μήπως είναι <laughs> γαλλικά του Λουξεμβούργου. Όχι είναι πολύ ωραία φωνή αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. <laughs> Στο τρία να συνεχίσω. Μα άκου το πρωτότυπο είναι στο μηδέν. Ναι, αλλά δεν είναι normal αυτό το πράγμα να ακούω άλλη γλώσσα στο 3. Να αρχίσω, να συνεχίσω. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Ως συνήθω, όπως ήθιστε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου τους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίας. Η ποσότητά τους είναι διαχειρίσιμη, 218. Φοβόμουν ότι θα είχαν κατατεθεί χίλιες και πάνω. Βέβαια διαπραγματεύτηκα με τους συναδέλφους για να καταλήξω στο μέγιστο δυνατό αριθμό συμβιβασμών και μία μορφή της έκθεσης που να μπορούν να τη δεχτούν οι περισσότεροι της Επιτροπής μας. Λέω αμέσως in medias res να αρχίσουμε να ομαδοποιούμε τις τροπολογίες κατά μεγάλα θέματα. Λοιπόν, καταρχήν μία πρόταση απόρριψης του κειμένου. Πρόταση η οποία στηρίζεται και από έναν συνάδελφο του ΕΛΚ και από έναν συνάδελφο των Σοσιαλιστών. Και αυτό δείχνει ότι η πρόταση της Κομισιόν ε, δημιουργεί πολλές αντιδράσεις. Κατανοώ τη σκέψη των δύο αυτών συναδέλφων και όσων το πρότειναν αυτό την διαγραφή δηλαδή, αλλά είναι αυτός ο ρόλος μας. Ομολογώ ότι έχω αμφιβολίες και θεωρώ φρονιμότερο να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις που να μπορούν να γίνουν δεκτές από το Συμβούλιο γιατί το να τα όλα έτσι βία νομίζω δεν θα βελτιώσει τα πράγματα εκτός αν πλειοψηφία συναδέλφων εδώ υποστηρίζει την πρόταση αυτή διαγραφής. Σε αυτή την περίπτωση φυσικά θα τη δεχτώ κι εγώ. Λοιπόν, άλλο είδος. Οι Πολωνοί συνάδελφοι προτείνουν ο, η φορολόγηση της εκπομπής διοξιδίου να είναι προαιρετική για κάθε κράτος μέλος. Η Κομισιόν λέει όμως ήδη να δοθεί παράταση της μεταβατικής περίοδου για, την, περίοδου για την εφαρμογή της φορολόγησης αυτής από τα καινούργια κράτη. Τώρα πρέπει γενικά να γίνει η προαιρετική φορολογία αυτή, δεν είμαι σίγουρη, αν και πάλι κατανοώ τη σκέψη των Πολωνών συναδέλφων. Έχω πάλι αμφιβολίες προς το παρόν τουλάχιστον γιατί δεν είναι τελειωτική η θέση μου. Αν γίνει όμως όλο το σύστημα προαιρετικό τότε δημιουργούμε νέους φραγμούς στην λειτουργία της έννοιας αγοράς που ήδη έχει πολλούς. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να τρευλωθεί η ισορροπία μέσα στην Ένωση αν ακολουθήσουμε αυτά που μας λένε οι Πολωνοί συνάδελφοι εφόσον θεωρούμε ότι είναι δικαιολογημένος ο φόρος αυτός, ας επιβληθεί παντού και μάλιστα με υποφερτό ποσοστό για από όλα τα κράτη-μέλη. Ίσως εδώ μπορεί να παίξουμε με τις διορίες και τις προθεσμίες της εφαρμογής, αλλά εσείς θα μου πείτε. μου πείτε. Τρίτον, για τον αναλογικό ή χαρακτήρα. Με χαρά βλέπω ότι πολλοί συνάδελφοι κατέθεσαν τροπολογίες με το ίδιο πνεύμα με το δικό μου, δηλαδή πολλοί ζητούν την κατάργηση των μηχανισμών αυτών που θα είχαν πολύ βαριές επιπτώσεις στην τιμή των καφουσίμων, ιδιαίτερα του ντίζελ. Και έπειτα και στο σύνολο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τις μεταφορές και στον πληθωρισμό. Να μην ξεχνάμε ότι από τότε που συζητάμε το θέμα η Ένωση βυθίστηκε στην κρίση. Η κακή αυτή, το κακό οικονομικό κλίμα, ίσως και πολύ κακό μάλιστα, μου δείχνει ότι σωστό είναι να μην ακολουθήσουμε την Κομισιόν επ' αυτού. Ο κύριος Λούτβικσον που είναι σκιώδης και σοσιαλιστής δεν συμφωνεί. Και καθώς είναι μεγάλη ομάδα και έχουν και αυτοί διαφορετικές απόψεις, νόμιζα ότι μόνο στο ΕΛΚ έχουμε διαφορετικές, αλλά έχουν και αυτοί, λοιπόν διαφωνεί και προτείνει να παραταθεί η προθεσμία στο 2018 αντί από το 18 στο 23 ή μάλλον από το 23 στο 28. Αλλιώς θα υπήρχαν αρνητικές επιπτώσεις πάνω στη λειτουργία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Θέλω όμως και εδώ να δω τι φρονούν οι περισσότεροι συνάδελφοι, η πλειοψηφία τους. Τέταρτον, και παραπλήσιον Διαπίστωσα ότι η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή δεν στηρίζεται εδώ από τα μέλη. Και νομίζω ότι σωστό είναι και αυτό. Η αυτόματη προσαρμογή από την Κομισιόν είναι κάτι που δε, με το οποίο δεν συμφωνούμε. Μερικοί μάλιστα βιαίως. Άλλοι θεωρούν ότι το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει και με ομοφωνία. Αλλά όπως ξέρετε το Συμβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτα αν δεν υπάρχει πρώτερη πρόταση της Κομισιόν. Έτσι γίνεται συνήθως. Πέμπτον. Οι εξαιρέσεις οι οποίες αφορούν πολλούς τομείς. Πρώτον, πολλοί συνάδελφοι ζητούν την κατάργηση της εξαίρεσης για τις θαλάσσιες και αεναέριες μεταφορές. Άλλοι λένε να μπει στο γενικότερο πλαίσιο εφαρμογής αυτό το μέτρο των εξαιρέσεων, άλλοι λένε να είναι προαιρετικές καθαρά. Εδώ θέλω η Κομισιόν να μας πει, σαφώς όμως, γιατί ήδη μίλησα στο διάδρομο με τον εκπρόσωπό της. Εγώ είχα καταλάβει ότι η συμπερίληψη των αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών δεν γίνεται νομικά λόγω της υπογραφής διεθνών συμβάσεων που έχουμε κάνει. Και μου λένε επίσης ότι δεν γίνεται νομικά για τις αεροπορικές μεταφορές συγκεκριμένα, αλλά ίσως λίγο περισσότερο για τις θαλάσσιες. Άλλοι συνάδελφοι λένε το αντίθετο. Δηλαδή αναφέρονται σε μία μελέτη αξιολόγησης από αυτές που κάνει τακτικά η Κομισιόν. Λες και το θέμα δεν είχε ακόμη λυθεί. Πριν τεθεί το θέμα πολιτικά, θα ήθελα να έχουμε την νομική απάντηση που μου τη δώσαν στο διάδρομο. Και πρέπει επίσης η Κομισιόν να πάρει κάποια θέση επίσημα για να είναι τα πράγματα σαφή. Άλλο παρόμοιο πρόβλημα, οι εξαιρέσει για εμπορική χρήση του ντίζελ μερικά λίγα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτό το δικαίωμα. Η πρόταση όμως της Κομισιόν είναι να καταργηθεί. Επ' αυτού έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες που ζητούν τη διατήρηση της εξαίρεσης αυτής. Για να είμαστε συνεπείς εγώ θα έλεγα μάλλον να καταργηθεί αλλά με σεβασμό βέβαια του αναλογικού χαρακτήρα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αναλογικότητα και μόνον μείνουν τα κατώτατα όρια, τα κατόφλια, τότε το θέμα της εξαίρεσης του τομέα αυτού, για εμπορική χρήση του ντίζελ δηλαδή, τότε γίνεται λιγότερο σημαντικό θέμα. Πρέπει να το ξαναδούμε λοιπόν και αυτό. Άλλο πρόβλημα, οι μη ορυκτές ενεργειακές πηγές και οι ανανεώσιμες. Και αυτό σημαντική πτυχή του ίδιου θέματος των εξαιρέσεων δηλαδή. Το θέμα είναι κάθε είδος ενεργείας θα το χειριστούμε ουδέτερα και ομοιόμορφα. Δηλαδή σύμφωνα με το πόσες εκπομπές διοξιδίου παράγει και πόση ενέργεια παράλληλα παράγει ή μήπως πρέπει να προβλέψουμε πιο διαφοροποιημένη αντιμετώπιση ανάλογα με άλλα κριτήρια που μπορεί και αυτά να είναι θεμητά. Για το υγροποιημένο αέριο, το φυσικό αέριο, ήδη πρότεινα μία διαφοροποιημένη αντιμετώπιση και ορισμένοι συνάδελφοι θέλουν να προχωρήσουν ακόμα παραπέρα. Το θέμα των βιοκαυσίμων επίσης συζητιέται από πολλούς συναδέλφους. Θα κάνω συνεννοήσεις για να δω πώς μπορώ να συνδυάσω αυτές τις απόψεις και να βρω κάτι το συνεπές, διότι η οδηγία που έχει σαν κύριο στόχο ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση των ειδών ενεργείας πρέπει να παραμείνει σε αυτό το πνεύμα έστω και αν αγκριθούν εξαιρέσεις όπου είναι όντως απαραίτητο. Τέταρτο γενικό θέμα για τις εξαιρέσεις πάλι, τέταρτη πτυχή. Οι εξαιρέσεις που χορηγούνται στη γεωργία και τη δασοκομεία κλπ. Η Κομισιόν προτείνει τέτοιες εξαιρέσεις, πρότεινε στο αρχικό της κείμενο, πολλές τροπολογίες όμως όπως και οι δικές μου την υποστηρίζουν αλλά ο σοσιαλιστής και ο θέλει η ρήτρα αυτή να έχει ορισμένους όρους και ο κύριος Λάμπερτς ο πράσινος ζητάει ίση αντιμετώπιση όλων των τομέων της οικονομίας. Πρέπει βέβαια να δούμε τι θα μας πει και στη γνωμοδότησή της η Επιτροπή Γεωργίας. Τελευταίο γενικό θέμα για τις εξαιρέσεις πάντα, το θέμα της οικιακής θέρμανσης. Δεν είναι απλό θέμα. Και πολλοί συνάδελφοι κατέθεσαν τροπολογίες που ζητούν την κατάργηση αυτής της εξαίρεσης με παράλληλη ίσως παράλληλους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων των πτωχοτέρων νοικοκυριών. Δεν θα ήμουν κατά εφόσον δεν αυξήσει αυτό την γραφειοκρατία να μην οικοδομήσουμε πολύπλοκους μηχανισμούς αναδιανομής απλώς και μόνο γιατί θέλουμε πιο σωστές τιμές. Πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε εδώ και μπορείτε να με πείσετε αν θέλετε και αν μπορείτε. Αυτά κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι είναι τα κύρια θέματα των τροπολογιών. Με μεγάλο ενδιαφέρον θέλω να ακούσω τους συναδέλφους διότι ο αριθμός των τροπολογιών και των συντακτών αυτών δεν ανταποκρίνεται απαραίτητο και στην πλειοψηφία των απόψεων των συναδέλφων. Θέλω λοιπόν να τα δω καλύτερα. Ποιοι ακριβώς πόσοι θέλουν περισσότερα από ό,τι πρότεινε η Κομισιόν και ποιοι θέλουν λιγότερα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι οι δικές μου θέσεις είναι αρκετά κεντρώες. Οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν τον Ιανουάριο μεταξύ μου και των σκιωδών και των συντακτών και ελπίζω ότι η Επιτροπή μας θα επιλέξει τελικά λογικά πράγματα υπέρ της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επίσης βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις για τα πυρηνικά από τον πράσινο σκιώδη. Δεν πρόκειται εδώ σε αυτή την έκθεση και πρόταση καθόλου για πυρηνικά. Αλλά υπάρχει τροπολογία που ζητάει να συμπεριληφθούν. Εδώ ερωτώ. Η παραγωγή ηλεκτρισμού από την πυρηνική ενέργεια δεν καλύπτεται ήδη από το τεστ. Νομίζω και αυτό πρέπει να το δούμε. Να, αυτά σε περίληψη. Ελπίζω όσοι δεν μπόρεσαν να διαβάσουν τις 218 τροπολογίες να πήραν κάποια ιδέα και σας ευχαριστώ για την παρασαχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στους κοιόδης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Λέει ο κ. Θα, μπορέσω, θα ήθελα να αναφέρω κάποιες από τις απόψεις μας και θα ήθελα να προσπαθήσω να αναφέρω και κάποια στοιχεία από αυτά που έθιξε η κυρία Λούλινγκ. Παρατηρώ εκ νέου ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ καλή. Έχει κάνει μια διεξοδική ανάλυση και εδράζεται επί μιας καλής, ισορροπημένης αξιολόγησης αντικτύπου. Θεωρεί ότι όλα λειτουργούν αρκετά καλά. Η οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας είναι κάτι απαραίτητο για μια αξιόπιστη ενεργειακή πολιτική. Η νομοθεσία που έχουμε τώρα ξεπεραστεί και χρειάζεται αναθεώρηση για να λειτουργεί σωστά. Χωρίς αναθεώρηση είμαι βέβαιος ότι δεν θα πετύχουμε τους στόχους του 2020. έχουμε ευθύνε στους ώμου μας. Και αυτό είναι κάτι που θα επηρεάσει και μελλοντικέ γενιές. Άρα έχουμε πάρα πολλή ε, δουλειά μπροστά μας. Θα πρέπει να κάνουμε κάποια σαφή βήματα, αλλά πρέπει να έχουμε και μια σφαιρική εικόνα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο. Πλαίσιο που θα πρέπει να κρατήσει κάποιες δεκαετίες. Η Πολωνική Προεδρία δεν κατόρθωσε να κρατήσει τη θέση της δυστυχώς και τα κράτη-μέλη θα κάνουν κάποιες αλλαγές απλώς όσον αφορά τη φορολόγηση. Η ιδανική προεδρία που πρόκειται να αναλάβει τα καθήκοντά της πρέπει να πετύχει πιο επικοδομητικά αποτέλεσματα. Το Κοινοβούλιο πρέπει να κινηθεί σχετικά γρήγορα. Πρέπει ε, έχουμε μια συγκεκριμένη θέση που θα στρέφεται και προς το μέλλον. Με επικοδομητικά σχόλια μπορούμε να κινηθούμε σωστά. Θα ήταν απαράδεκτο αν καθυστερήσουμε περαιτέρω. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε και να δούμε τι θα συμβεί στο Συμβούλιο. Πρέπει να εισακουστούν οι απόψεις μας και για να γίνει αυτό θα πρέπει να εκφραστούμε έγκαιρα. Βλέποντας τις προτινόμενες τροπολογίες Πιστεύω ότι πρέπει να επεξεργαστούμε και να εξετάσουμε σοβαρά πέντε τομείς στις διαπραγματεύσεις. Καταρχάς, ακόμα και τα στέρεα βιοκαύσιμα θεωρείται θα πρέπει να φορολογηθούν. Ανεξάρτητα αν είναι βιώσιμα ή όχι. Δεν μπορούμε από πλευρά φορολογίας τα στερεά βιοκαύσιμα που δεν είναι βιώσιμα ε, να βρίσκονται σε προνομιούχα ε, θέση. Αυτό για μένα είναι αυταπόδεικτο. Ταυτόχρονα γεγονός είναι ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια όσον αφορά τα στέρεα βιοκαύσιμα. Ποια είναι τα κριτήρια βιωσιμότητας, Φερρυπίν. Ε, χρειάστηκε καιρός για να καταλήξουμε σε κάποιες ιδέες. Πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια κριτήρια που θα μπορούν να εφαρμόζονται το ταχύτερο δυνατόν στα πλαίσια της παρούσης οδηγίας. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτή την οδηγία είναι να μεταφέρουμε απλώς τα ίδια κριτήρια για τα στέρεα βιοκαύσιμα ε, που να είναι παρόμοια με τα άλλα βιοκαύσιμα. Η αρχή της βιωσιμότητας διαφέρει κατά κατηγορία. Γενική πολιτική δεν θα λειτουργούσε. Η αρχή της ουδετερότητας είναι πολύ σημαντικό θέμα. Κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να απαλλαγούμε από αυτό το κριτήριο. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Χρειαζόμαστε πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Είναι λογικό καταρχήν να αποφασίσουμε ότι κάθε καύσιμο που χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό να φορολογείται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι δίκαιο και δημιουργεί και προβλέψιμες συνθήκες για ισότιμο ανταγωνισμό. Αν δεν το δούμε τόσο ολιστικά και το δούμε πιο βραχυπρόθεσμα το θέμα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα προβλήματα. Η καλύτερη λύση είναι να πάρουμε την ουσία από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά να εξετάσουμε εκ του σύνεγγυης κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά την σταδιακή εφαρμογή και την περίοδο σταδικής εφαρμογής. Υπάρχουν επιχειρήματα που είναι υπέρ μεγαλύτερας περίοδου προσαρμογής. Τρίτον, σε διάφορους τομείς υπάρχει επιθυμία να διατηρηθούν ε, οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα για το εμπορικό ντίζελ. Πέντε χώρες μόνο χρησιμοποιούν μειωμένη φορολόγηση του καυσίμου αυτού. Είναι περιορισμένο φαινόμενο μπορώ να συζητήσω προφανώς κάποια σταδιακή εξάλληψη βραχυπρόθεσμα των κανόνων για το εμπορικό ντίζελ. Αλλά αυτή η παράμετρος δεν πρέπει να μείνει για πολύ περισσότερο εντός του νόμου. Τέταρτον, ε, αυτή η αναπροσαρμογή, η τιμαριθμική, ε, είναι ταμπού σε κάποιες χώρες. Εκεί στις χώρες που χρησιμοποιείται μια προσαρμογή, ε, τη μαριθμική της φορολόγηση των καυσίμων, δουλεύει καλά. Έχουμε τέτοια προσαρμογή στη Σουηδία για το διοξείδιο του άνθρακα. χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Αυτή η αναπροσαρμογή είναι καλός αποτελεσματικός τρόπος για να μην υπονομεύονται οι φορολογικοί συντελεστές. Το έχει σκεφτεί το θέμα ήδη και το έχει αναφέρει στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να προχωρήσουμε περισσότερο στο θέμα αυτό και να καταλήξουμε στο σωστό μηχανισμό. Να μπορέσουμε να συσχετίσουμε τα ελάχιστα επίπεδα ε, μονοξιδίου του άνθρακα με τη γενικότερη φορολόγηση των εκπομπών. Θέλουμε να όσον αφορά το εμπόριο ρήπων να επικρατούν ε, δίκαιες συνθήκες. Πρέπει να απαλλαγούμε επίσης από την υποχρεωτική εξαίρεση της φορολόγησης αερομεταφορών και θαλασσίων μεταφορών να γίνει ε, εθελοντική η εξαίρεση. Η απαγόρευση της φορολόγησης δεν δικαιολογείται από το διεθνές δίκαιο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν μέτρα που θα πρασινίσουν κατά κάποιο τρόπο τη χρήση ενέργειας. Ε, πρέπει να εξετάσουμε διεξοδικότητα τις λεπτομέρειες στις μελλοντικέ συζητήσει. Εγώ είμαι ανοιχτό. Χρειάζεται γενική θεώρηση των πραγμάτων. Θέλουμε να υπάρχει ευρία υποστήριξη Θέλουμε να τροφοδοτήσουμε το Συμβούλιο με τι απόψει μα, να κινηθούμε σωστή κατεύθυνση. Αυτέ είναι κάποιε από τι απόψει μα και προσβλέπουμε σε μελλοντικέ επικοδομητικέ συζητήσει και μέσω συζητήσεων να βρούμε κοινέ λύσει. Διότι θα είναι σημαντικό να αναθεωρηθεί η οδηγία για τη φορολόγηση των ενεργειακών πηγών. Δεν είναι ένα απλό θέμα αναθεώρησης. Μιλάμε για εξυγχρονισμό της νομοθεσίας. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ που είναι το λόγο και ευχαριστώ και την κυρία Λούλινγκ που έκανε μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση και ελπίζω να βρούμε κάποιες λύσεις με όλες τις ομάδες του Κοινοβουλίου και με όλους τους κοιόδης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και Πρόεδρος. Ο Φίλιπ έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστώ τον εισηγητή την εισηγήτρια συγκεκριμένα για το, την εργασία της. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και έχοντας αναδειφίσει τις τροπολογίες από τα διάφορα πολιτικά κόμματα βλέπω ότι υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει. Γιατί οι θέσεις των μεν και των δε φαίνεται να αποκλίνουν σημαντικά. Κάποιες γενικές αρχές θα ήθελα να εδραιώσω εδώ. Ως φιλελεύθεροι εμείς είμαστε υπέρ μιας μετατόπισης προς πιο πράσινη μορφή φορολογίας και την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους για τα ενεργειακά προϊόντα και ιδιαίτερα για τον ηλεκτρισμό. Είναι σημαντικό επίσης να εξασφαλίσουμε ισοτιμία ανταγωνισμού για όλα τα προϊόντα. Μιλάμε για μια φορολογία η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται με έναν τρόπο που είναι τεχνολογικά ουδέτερος. Επίσης θα πρέπει να καταστεί δυνατό για μας να δώσουμε την ευκαιρία σε νέες τεχνολογίες, τεχνολογίες που μπορεί να μην τις γνωρίζουμε καθόλου αυτή τη στιγμή, να καλυφθούν από αυτή την φορολογία. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω την πρόταση της Κομισιόν, τις δύο κύριες αρχές της πρότασης της Κομισιόν συγκεκριμένα, ένα διπλό στάδιο φορολογίας για το διοξείδιο του άνθρακος για να πετύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους και δεύτερον ένα γενικό φόρο κατανάλωσης που έχει να κάνει με το ενεργειακό περιεχόμενο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα μπορέσει να αυξήσει την αποδοτικότητα της χρήσης της ενέργειας. Είναι πολλά μέλη του Κοινοβουλίου που θέλουν να κάνουν προαιρετικό το κομμάτι που έχει να κάνει με τη φορολόγηση για το διοξείδιο του άνθρακος. Άλλοι όμως όπως εγώ θέλουν να το κάνουν δεσμευτικό και υποχρεωτικό. Θέλουμε να εξυγχρονίσουμε την οικονομία μας, θέλουμε να έχουμε πρασινότερη οικονομία και το στοιχείο του διοξείδου του είναι βασικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η αρχή της αναλογικότητας που υπενθύμησε η κυρία Λούλινγκ. Γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το τι σημαίνει αναλογικότητα. Αν θέλουμε να έχουμε ισοτιμία αναγωνισμού μεταξύ διαφορετικών φορέων ενέργειας, αυτό είναι ουσιώδες. Δεν μπορείτε να δώσετε προτεραιότητα σε μία μορφή ενέργειας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή της αναλογικότητας. Είδαμε και ακούσαμε παραδείγματα αναλογικότητος στην πράξη. Δεν πρέπει αυτό να οδηγήσει κατά ανάγκη και νομοτελειακά σε αύξηση των τιμών. Είναι απαραίτητο να έχουμε και μια περίοδο σταδιακής προσαρμογής. Πρέπει να σκεφτούμε και τον κύκλο επενδύσεων σε διάφορους τομείς και νομίζω θα είναι πάρα πολύ λογικό να έχουμε μεταβατικές περιόδους για να μπορέσουν και οι καταναλωτές και η παραγωγή ενέργειας να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα κατάσταση που επιθυμούμε να εισαγάγουμε. Είναι σημαντική λοιπόν και η επικουρικότητα. Πρέπει να βρούμε εφάνταστες λύσεις ώστε να καταλήξουμε σε μια σωστή θέση για τα ζητήματα αυτά. Υπάρχουν και άλλα σημεία τα οποία ανέφερε η κυρία Λούλινγκ. Ίσως ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτή τη στιγμή είναι η αυτόματη αναπροσαρμογή για, την, ε, για το φόρο κατανάλωσης στους καταναλωτές. Εδώ υπάρχουν κάποια προβλήματα με τον αυτόματο χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα επικίνδυνο προηγούμενο ότι όλες οι μορφές ε, φορολογίας θα αντιμετωπίζονται με τον τρόπο αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε και άλλες ε, εφάνταστες λύσεις για την αναπροσαρμογή, να μην είναι αυτόματη. Δεν συμφωνώ και με την εξαίρεση για νοικοκυριά για κοινωνικούς λόγους. Νομίζω ότι όλοι οι τομείς είτε είναι καταναλωτικοί είτε είναι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν σαφή μηνύματα για να μπορέσουν να σχεδιάσουν καλύτερα για το μέλλον. Μπορεί να υπάρχει μια αντισταθμιστική πληρωμή για κοινωνικούς λόγους για αυτά τα θέματα, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση για την αποδοτικότητα της ενέργειας. Και έχουμε και τους τομείς που είναι έντασης ενέργειας. Εκεί δεν πρέπει να έχουμε μία επικάλυψη με το σύστημα ETS των εκπομπών εμποριών, των εμποριών εκπομπών. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν απουσία διπλής φορολόγησης και να δώσουμε στη βιομηχανία το χρόνο να προσαρμοστεί. Πρέπει επίσης να δούμε και το διεθνές πλαίσιο όπως ανέφεραν ορισμένοι συνάδελφοι το μέλλον δεν είναι πάντα τόσο λαμπρό και γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε τις μεταβατικές περιόδους και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει συνεκτικότητα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο φορολογούμε και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το πλαίσιο που θέλουμε να αναπτύξουμε είναι πραγματικά σφιχτό και θα εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχουν σημεία σημαντικά που υπάρχει διαφορά απόψεων για τις εξαιρέσεις σε ορισμένου τομεί. Και υπάρχουν πτυχέ που αναφέρθηκαν προηγουμένω. Αλλά σα λέω και πάλι, μια συνεκτική και συνεπής προσέγγιση είναι πάρα πολύ σημαντική και μπορούμε μαζί με του κοιόδης συζητητές να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποιε συμβαστικέ λύσει, γιατί αυτό είναι και ο στόχο μα. Είναι ένα πάρα πολύ πολιτικά ευαίσθητα θέμα στο Συμβούλιο και στην πράξη έχει μπλοκαριστεί. Από την πλευρά του Κοινοβουλίου όμω θα πρέπει να το δούμε αυτό σαν μια ευκαιρία. Δεν πρέπει να υστερήσουμε του Συμβουλίου, πρέπει να παίξουμε ηγετικό ρόλο να κάνουμε απόλυτα σαφές ποια είναι η θέση μας και να προωθήσουμε τις απόψεις μας και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επηρεάσουμε και τη γραμμή που θα υιοθετήσει στο Συμβούλιο. Προσβλέπω λοιπόν σε μια σειρά επικοδομητικών συζητήσεων τον Ιανουάριο. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το θέμα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία να τολμήσουμε και να βοηθήσουμε τους πολίτες μας να προχωρήσουμε προς την πράσινη οικονομία. Ευχαριστώ, Λεκή Πρόεδρο. Κάποιος από τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστές. Όχι. Ο Φιλίπ. Θα ακούσεις πάνω ιστορία από τους δύο φίλοι που σήμερα. Πρέπει να πω ότι πράγματι δεν θα επαναλάβω αυτό που είπε ο Φιλίπ ε, μόλις τώρα. Πολύ καλή πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Κάποια φορά κανείς θεωρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν τον αρχιτέκτονα της λιτότητας, αλλά μπορεί να βλέπει και μακριά στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και, εφόσον, και ότι προσπαθούν αυτή τη φορά να μας βήξουν προς τα μπρος. Και δεν θα πρέπει να χαλάμε την απόλαυσή μας, μάλλον μην χάσουμε την ευκαιρία μάλλον. Λοιπόν, τούτου λεχθέντος θα, θα πρέπει να δούμε ότι έχουμε μεγάλη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε, άρα δεν θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα πλευρά φορολόγηση ή να καθυστερήσουμε ή να ακυρώσουμε την πρωτοβουλία διατείνονται κάποιοι όπω ο Λάγκεν και ο Γκέπελ από πλευρά S&D και ΕΛΚ. Αυτό θέλουν να πιστέψουμε. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι. Ότι πρέπει να διαβάσουμε ξανά την έκθεση Stern ε, χρονολογείται από πέντε χρόνια. Εκεί παρουσιαζόταν η οικονομική συνέπεια της αλλαγής του κλίματος. Και η οικονομική συνέπεια δεν πρέπει να υποτιμάται. Αν όλοι σε εσάς σοβαροί και θέλετε να ανθίσει η οικονομία μας, δεν μπορείτε να αρνηθείτε την ανάγκη καταπολεμήσεως αλλαγής του κλίματος. Διότι μπορεί αυτό να έχει τεράστιο αντίκτυπο οικονομικό και είναι θέμα ζωής και θανάτου, όχι κάπου αλλού στον πλανήτη μόνο, αλλά και στην Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή είναι κρίση αυτή θα περιμένει η αλλαγή του κλίματος. Η αλλαγή του κλίματος δεν περιμένει και σας παροτρύνω να ξαναδιαβάσετε τα συμπεράσματα του IPCC. Αν θέλουμε να σώσουμε τις οικονομίες μας, καλό θα είναι να ασχοληθούμε με την αλλαγή του κλίματος. Αλλά και βραχυπρόθεσμα θα ήταν καλό για την οικονομία να κάνουμε αυτό που είπε ο Φιλίπ. Να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους τομείς, κυρίως όσον αφορά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμες μεταφορές, ενέργεια για στέγαση κλπ. Να μην χάσουμε την ευκαιρία να τους δώσουμε την οικονομική ευκαιρία που τους αξίζει. Και τώρα οι αρνητικές επιδοτήσεις που δίνονται στα ορυκτά καύσιμα τις εμποδίζουν αυτές τις ενέργειες. Το status quo είναι κακό για την οικονομία μας. Αυτό που είναι καλό για την οικονομία είναι να προχωράμε με ενεργειακό φόρο, λογικότερο. Έχουμε για μια φορά μια πρόταση που καταλαβαίνουμε σε ποια λογική στηρίζεται. Είναι συνέπειες του διεξιδίου του άνθρακου στο ενεργειακό περιεχόμενο. Ε, ηλίου φαϊνότερο το περιεχόμενο. Καμία από τις δύο πτυχές κατά την άποψή μου δεν πρέπει να είναι προαιρετική και όσο πιο γρήγορα φτάσουμε στο αποτέλεσμα θέλουμε το καλύτερο. Και δεύτερον, αυτοί που διατείνονται ότι χρειαζόμαστε χρόνο για την αλλαγή, συμφωνώ, συμφωνώ με αυτό που λένε. Η αλλαγή των μορφών φορολόγηση δεν είναι κάτι που γίνεται μία ανοιχτή. Όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι τόσο ανόητη να προτείνει μια τέτοια αλλαγή σε μία νύχτα. Αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να ξεκινήσουμε την αλλαγή το 2023, σε 12 χρόνια από τώρα δηλαδή. 2023. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη θα υπάρχουν ακόμα τότε, ελπίζω, αλλά είναι σχεδόν άλλο αιώνα. Δεν είναι ότι δεν έχουν χρόνο να προσαρμοστούν οι βιομηχανία και οι καταναλωτές. Πιστεύουμε ότι οι μεταβατικές περίοδοι και το σχέδιο το μεταβατικό πιθανότατα ήδη υπολείπονται των όσων θα μας υποχρεώσει να κάνουμε η φύση. Υποτιμούμε και τον αντίκτυπο που θα έχει η οικονομία και το κλίμα στην Ευρώπη. Άρα αυτοί που θέλουν έτσι περαιτέρω καθυστέρηση ε, σφάλουν. Αν το κάνουμε αυτό, η Ευρώπη δεν θα είναι ανταγωνιστική. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μην κάνουμε αλλαγή. Κάποιοι το S&D και το ΕΛΚ Πώς θέλετε να γίνει η χρηματοδότηση, αν δεν θέλετε να φορολογήσουμε το χρηματοδοτικό τομέα. Άλλοι λένε να μην αυξήσουμε τους ενεργειακούς φόρους. Να μην βάλουμε φόρο στο ένα ή στο άλλο, σε τι καταλήγουμε. Φορολογούμε το εισόδημα. Φόρο εισοδήματο. Αυτό είναι το μόνο που μένει να φορολογηθεί. Και όλοι λέμε ότι δεν πρέπει να φορολογήσουμε των εργαζομένων το εισόδημα. Πού θα βρούμε πόρους όμως. Αυτή η οδηγία για τον ενεργειακό φόρο, και εδώ διαφωνώ με τον Φιλίπ, πιθανότατα θα καταλήξει σε υψηλότερου φόρου επί τη ενέργεια. Αλλά, και εδώ είναι η αντιστάθμιση, αυτό θα έπρεπε να μεταφραστεί σε χαμηλότερη ε, φορολόγηση εσόδων των εργαζομένων. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ούτω ώστε να γίνει η απασχόληση πιο ελκυστική και για του εργοδότε και τους εργαζόμενους. Και αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να αναφέρω και κάποια άλλα θέματα. Η αναπροσαρμογή. Καταλαβαίνω την ησυχία σου, Φιλίπ. Δεν θέλει η αναπροσαρμογή να γίνει ο γενικό κανόνα. Εδώ, στον τομέα τη ενέργεια, η αναπροσαρμογή δικαιολογείται λόγω τη αλλαγή του κλίματο. Διότι γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε αύξηση τη τιμή του διοξιδίου του άνθρακο, αν θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακος. Και θα πρέπει να φτάσουν στο υψηλότερο σημείο της καμπύλης τώρα και να μειωθούν στο μέτρο του δυνατού του 2050. Αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να προτείνουμε να σχεδιάσουμε την τροχιά μας. Και εδώ η αναπροσαρμογή είναι κάτι λογικό, διότι υπάρχει ένας φυσικός περιορισμός που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Δεν είναι ότι ξέρουμε ότι θα ψηθούν οι τιμές και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα πάρουμε περισσότερα χρήματα. Δεν είναι αυτό. Θέλουμε να αποθαρρύνουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, ούτως ώστε να ακολουθήσουμε τη σωστή τροχιά. Και εδώ χρειάζεται η αναπροσαρμογή. Οι εξαιρέσει κάθε φορά που αναφέρεται κανείς στη φορολόγηση κάποιος θα πει καλός αλλά όχι εμένα. Εγώ θέλω να εξαιρεθώ. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχει κάποιο σχήμα, πρέπει να ξεφύγουμε. Το νόημα της ανανεωμένης φορολογίας είναι ότι πλήττει την κατανάλωση ενέργεια σε εκπομπέ διοξιδίου στο άνθρακο. Πρέπει ε, να έχει πυγμή. Αν δεν έχει πυγμή η φορολόγηση, δεν θα αλλάξει τι συμπεριφορέ. Και συμφωνώ με αυτό που είπε ο Φιλίπ. Και κοινωνικό τομέα θα πρέπει να εξαιρεθεί, κοινωνική πολιτική. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε σαν πανάκια ε, έναν φόρο. Ένας ενιαίος φόρος δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Για να μειωθούν οι κοινωνικές συνέπειες των υψηλότερων ενεργειακών τιμών ε, μπορούμε να φροντίσουμε τι θα γίνει με την φορολόγηση εισοδήματο. Και για τα ευάλωτα νοικοκυριά μπορούμε να μειώσουμε τη φορολόγηση. Έχουμε διάφορα εργαλεία φορολογικά που χρησιμοποιήσουμε. Και δεν ταιριάζει ένα μέσο για όλους τους σκοπούς. Αυτά έχω να πω ε, και προσβλέπω στον Ιανουάριο σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ντανούτα Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την κυρία Λούλιν για την πολύ βαθιά ανάλυση της σε σχέση με αυτά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω να την ευχαριστήσω για την κατανόηση που έδειξε για τις τροπολογίες που μπορέσαμε να παρουσιάσουμε για την φορολογία διοξιδίου του άνθρακος. Ένας υποχρεωτικός φόρος διοξιδίου του άνθρακος δεν μπορεί βέβαια να εφαρμοστεί χωρίς να υπάρχει μια βαθιά ανάλυση. Και επομένως θα πρέπει να υπάρξει και μια ανάλυση του πώς αυτό θα επηρεάσει την κατανάλωση ενέργειας. Νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει να προχωρήσουμε προς ένα καταρχήν προαιρετικό φόρο διοξιδίου του άνθρακος και ο υποχρεωτικός φόρος διοξιδίου του άνθρακος θα πρέπει να αναβληθεί για ένα μεταγενέστερο χρονικό ορίζοντα όταν υπάρχει και πλήρης ανάλυση και στα κρατημέλη αλλά και στη σύνολη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος. Η Αστρίδα. Κάτι γράφει σε Αστρίδα, αλλά νομίζω ότι μπορείς να έχεις το λόγο που θέλεις. Τελειώσατε όλοι. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Όχι. Όχι. Η Κομισιόν θέλει να πει κάτι σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ναι, ναι, παρακαλώ. Η Αστή θέλει να θέσει κάποια ερωτήματα ούτως ή άλλως, οπότε η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει στη συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λούλιν και τους σκιώδεις εισηγητές για την γενικά υποστηρικτική συμβολή τους στην έκθεση αυτή και για τις τροπολογίες τους. Είναι πολλές βέβαια οι τροπολογίες. Από την πλευρά της Κομισιόν προσπαθήσαμε να τις ομοδοποιήσουμε <clears throat> και έτσι έχουμε κατατάξει σε περίπου 40 κατηγορίες. Δεν πρόκειται να τις απαριθμίσω βέβαια. Απλώς περιορίζομαι σε ορισμένα κέρια θέματα και κυρίως αυτό το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για την κυρία Λούλινγκ που αφορά τις διεθνείς αεροπορικές και ναυτιλιακές συγκοινωνίες που πράγματι πρέπει να αντιμετωπιστούν χωριστά. Αν δούμε τον τομέα της αεροπορίας, ο τομέας αυτός θα περιληφθεί στο σύστημα εμπορίας εκπομπών από το 2012. Και ακολουθώντας τη λογική της πρότασής μας, οι οικονομικοί τομείς που υπόκεινται στο σύστημα εμπορία εκπομπών δεν πρέπει να υπόκεινται στην οδηγία φορολογίας τη ενέργεια. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι ήταν σωστό και πρέπει να μην προτείνουμε περαιτέρω φορολογία του τομέα αεροπορικών μεταφορών σε αυτό το νομοθέτημα. Επίσης, όπως ελέγχθη, είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του τομέα της ε, των αεροπορικών συγκοινωνιών συμμετέχει σε διάφορες διεθνείς συμβάσεις όπως είναι η σύμβαση του Σικάγου. Επομένως, ό,τι και να συμπεριλάβουμε εδώ θα περιλαμβάνει μόνο ένα περιορισμένο τμήμα της διεθνούς των αεροπορικών διακινήσεων, δηλαδή μεταξύ 100 μερών συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή όλες αυτές οι διεθνείς συμβάσεις είναι έτοιμες για επαναδιαπραγμάτευση, στο άμεσο μέλλον, αυτό θα υποβάθμιζε την ε, διαπραγματευτική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου. Και ουσιαστικά δεν θα άλλαζε πάρα πολύ τη συνολική φορολογία των μεταφορών. Διαφορετικά είναι τα πράγματα για τις ναυτικές μεταφορές και εδώ υπάρχουν συμβάσεις για τους εσωτερικούς ε, υδάτινους δρόμους, η λεγόμενη σύμβαση του Μανχάιμ, όπου προβλέπονται ορισμένε εξαιρέσεις αλλά για να αλλάξουμε τους κανόνες εδώ υπάρχει πολύ περισσότερο περιθώριο από στην αεροπορικό, στον αεροπορικό κλάδο. Γι' αυτό η Κομισιόν, οι υπηρεσίε τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, κάνουν τώρα μία έκθεση, μία ανάλυση αντικτύπου σε σχέση με τις συνέπειες οι οποίε θα μπορούσαν να προκύψουν από μία αλλαγή των κανόνων. Περιμένουμε μέσα στον επόμενο χρόνο να έχουμε τα στοιχεία από αυτή την ανάλυση, επί τη βάση των οποίων εξελίξεων και αναλύσεων θα μπορέσουμε να προτείνουμε τε... αλλαγές στο πλαίσιο αυτό. Και επίσης συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας και πιστεύουμε ότι θα ήταν λογικό να περιμένουμε για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων αυτών. Χωρίς τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, τις 219 τροπολογίες, κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Κάποιες ε, τροπολογίες θέλαν να διευρύνουν την εμβέλεια εφαρμογής της πρότασης της Κομισιόν, φορολογία αυτοκίνητων οχημάτων, ταξινόμουσια οχημάτων, ε, προσδιορισμό των πόρων που θα προκύψουν αυτή η φορολογία, συμπερίληψη πυρηνική ενέργεια κτλ. Όλα αυτά καταρχήν δεν υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο της τωρινής οδηγίας ενέργειας, οπότε θα ήταν δύσκολο για την Κομισιόν να προτείνει αλλαγές προς την κατεύθυνση αυτή. Απιπλέον σε ό,τι αφορά την, τα φορολογία οχημάτων και τον προσδιορισμό, αυτό ουσιαστικά παραβιάζει την αρχή της επικορικότητας που δίνει υψηλή ε, υπευθυνότητα στα ευθύνη στα μελη για να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές. Το να μην υπάρχει το στοιχείο διοξιδίου του άνθρωπου στην πρόταση αυτή, κατά την άποψή μας, θα καταργούσε ένα από τα βασικά στοιχεία αυτής της μεταρρύθμισης και θα απογύμνωνε αυτό το περιεχόμενο της πρότασής μας. Πρέπει να τονίσουμε και πάλι ότι υπήρξε μια πραγματική εντολή που δόθηκε από τα άλλα θεσμικά όργανα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2008 να αλλάξει η φορολογία της ενέργειας για να, ενέργειας για να συμπεριλάβει και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για την γεωργία, δεν ξέρω σε πόσο βαθμό λεπτομέρειες θέλετε να προχωρήσω έχω να ακούσω την εισηγήτρια και στις 4.30 έρχεται ο Μάριο Ντράγκη. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε λίγο πιο σύντομος. Έχω τουλάχιστον λίγο χρόνο. Μπορώ να αναφερθώ σε μερικές από τις πιο σημαντικές ομάδες τροπολογιών. Υπήρχε συζήτηση για το θέμα των τομέων γεωργίας, ε, παραγωγής ε, φρούτων και λαχανικών, υδρο, υδατοκαλλιεργειών κτλ. Δεν θεωρούνται ότι είναι βασικές πηγές διοξιδίου του άνθρακος, εκτός αν υπάρξει κάποια, ε, κάποια ένδειξη ότι υπάρχει ο κίνδυνος μετακίνηση αυτών των επιχειρήσεων, λεγόμενης διαρροής άνθρακος στο τμήμα που έχει να κάνει με την φορολογία της ενέργειας υπάρχει πάντα δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να δώσουν εξαιρέσει εάν υπάρχει και κάποιο αντιστάθμισμα στο περιβάλλον και υπάρχει κάποια λογική που είναι συνεκτική και συνάδει για την ενεργειακή φορολογία. Τέτοιου είδους προτιμησιακές ε, μεταχειρήσεις όπως είναι το αγροτικό ντίζελ μπορούν να διατηρηθούν. Επίσης προτάθηκε από ορισμένου ότι άλλα αέρια του θερμοκηπίου ή άλλες ε, πηγές άχθους, εξτernalities δηλαδή, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτές. Αυτό το εξετάζουμε στην ε, ανάλυση η οποία έγινε πριν από τη διατύπωση αυτής της πρότασης, externalities του διοξιδίου του άνθρακος είναι οι μόνες εκπομπές που είναι πραγματικά διαμεθοριακές και είναι σαφώς συνδεόμενες με καύσιμα και χρήση τεχνολογίας. Γι' αυτό μια επέκταση σε άλλες πηγές εξωτερικών, εξωτερικού άχθους δεν θα ήταν πρόσφορη. Σταματάω λοιπόν εδώ. <clears throat> Σίγουρα. Λοιπόν, θα τα διαβιβάσω με αυτά, αλλά πρέπει να φύγω μερικά λεπτά, ούτως ώστε η συγγήτρια να πάρει το λόγο. Ε, για έχει το λόγο, η συγγήτρια. Ναι, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς δεν είμαι πιο εν, ενήμερη από ό,τι πριν, διότι διαπιστώνω πάντα ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις απόψεων. Διαπίστωσα ότι όσον αφορά την αναλογικότητα έχουμε πραγματικά σημαντικές διαφορές. Διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των απόψεων εκείνων των συναδέλφων που υπέβαλαν τροπολογίες. Πιστεύω ότι οι σκιώδεις θα είχαν την τάση να είναι περισσότερο υπέρ με μεγάλη αύξηση των προθεσμιών προφανώς. Το σημαντικότερο είναι ότι εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας είπε ότι τι δεν συμπεριλαμβάνεται. Και ελπίζω ότι οι συντάκτε των τροπολογιών κατανοούν ότι δεν πρέπει να μιλάμε για τον τομέα των αρμεταφορών διότι υπάρχει μια σύμβαση και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα τώρα όσον αφορά τη σύμβαση αυτή για τις αλλαγές μεταφορές και τη σχετική σύμβαση θα πρέπει να περιμένουμε την μελέτη αντικτύπων μέχρι ότου αλλάξουμε κάτι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προτείνει να εξαιρεθούν αυτοί οι δύο τομείς. Έλαβα γνώση και του ότι δεν πρέπει να μιλάμε στις τροπολογίες μας για φόρους που δεν έχουν καμία σχέση με ενεργειακό φόρο όπως είναι ο φόρος των αυτοκινήτων. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Εξίσου σημαντικό είναι αυτή την ιδιαίτερη αντιμετώπιση να την επιφυλάξουμε και για τη Γεωργία. Υπάρχουν αποκλήσεις απόψεων επίσης όσον αφορά την αναπροσαρμογή, την αναλογικότητα. Δεν μιλήσαμε για, την πυρηνική, ε, για τον πυρηνικό τομέα, διότι πιστεύω δεν πρέπει να συζητηθεί εδώ. Διαπίστωσα την απόσταση αυτή που υπάρχει μεταξύ των απόψεων. Δυστυχώς μάλλον δυστυχώς δεν ήταν εδώ κάποιος από τους συναδέλφους που είναι κατά της προτάσεως και που υπέβαλαν τροπολογίες που ξεπερνούν τις προτάσεις συναδέλφων τους της ομάδας. Είναι αυτοί που δεν θέλουν να προχωρήσουν τόσο πολύ όσον αφορά τη φορολόγηση και μάλιστα δεν θέλουν να προχωρήσουμε γρήγορα. Εγώ προτείνω τον Ιανουάριο να ξεκινήσω συζητήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές και με τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες που ακολουθούν εντελώς διαφορετική νοοτροπία να δούμε ποιες είναι οι απόψεις των σκιωδών και ελπίζω να καταλήξω στο να προτείνω κάποιες τροπολογίες που θα μπορούν να υποστηριχθούν από την πλειοψηφία. Γνωρίζω τι συμβαίνει στο Συμβούλιο. Ήρθα σε επαφή και με την Δανέζικη Προεδρία. Πρέπει να σε επαφή μάλλον με την Δανέζικη Προεδρία. θα προσπαθήσω να δω κατά πόσο μπορεί να διαμορφωθεί μια πλειοψηφία επί κάποιων συμβαστικών προτάσεων. Να βρούμε ισορροπία μεταξύ εκείνων που θέλουν να προχωρήσουν πιο πέρα από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκείνων που δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Θα το σκεφτώ κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε να ψηφίσουμε στις 28 Φεβρουαρίου και να πάμε στην πρώτη ολομέλεια του Απριλίου, όπως είπε και η Άστριτ, Χρειάζεται κάποιο χρόνο για να συζητήσει το θέμα με συναδέλφους. Αυτό είναι το παρόν χρονοδιάγραμμα. Τώρα. Πάμε τώρα στο σημείο 5 που αφορά το διάλογο με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αν μου επιτρέπετε θα πάω να δω και πού βρίσκεται ο κύριος Τρέγκη. Okay, time over Πέρασε η ώρα των φωτογραφιών. Πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε στο διάλογο περί νομισματικών. Για τα μέλη που δεν ήταν εδώ προηγουμένως όταν έκανε τι ανακοινώσει Προέδρου, πρέπει να σας πω ότι έγινε τη επίσκεψή μας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόσφατα και είχαμε τη δυνατότητα ανεπισήμων συνομιλιών και επαφών με τον νέο πρόεδρο μας. Καλωσορίζω με τα χαρά τον Μάριο στην πρώτη του συμμετοχή στον Ουσβατικό Διάλογο. Όπως ξέρουμε θα έρχεται εδώ τακτικά, αρκετά τακτικά και σαν πρόεδρος της ΕΚΤ και σαν πρόεδρος του, Συμβουλίου για τον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Συστημικό Κίνδυνο. Εξακολουθούμε να διαχωρίζουμε αυτά τα είδη των διαλόγων διότι διαφορετικά θα μπορούσαμε να καλύψουμε τα πάντα σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλιά σας ε, στους Financial Times. Μάλλον έκαναν πολύ ενδιαφέροντες τίτλους ε, από αυτά που είπες που δεν ήταν τόσο ενδιαφέροντα αλλά τα έκαναν ακόμη πιο ενδιαφέροντα σαν τίτλους. Σου δίνω το λόγο για να μας συνοψίσεις τη θέση στην οποία βρισκόμαστε και μετά θα ακολουθήσει η περίοδος των ερωταπαντήσεων. Έχεις το λόγο Μάριο και καλώς ήρθες. Ευχαριστώ Σάρν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αγαπητά αξιότιμα μέλη. Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά να συμμετέχω για πρώτη φορά σαν Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, σε αυτή την ακρόαση. Οι τριμηνίες αυτές ακροάσεις στην ΕΚΟΝ είναι ακρογωνίας λήθους για επικοδομητική σχέση μεταξύ των δύο θεσμών μας. Αυτή η ανταλλαγή έγινε εδώ και μερικούς, μερικές εβδομάδες μετά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που ελήφθησαν και από το Συμβούλιο των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από τους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο η συζήτησή μας υπόσχεται να είναι ιδιαίτερος πλούσια και καρποφόρα. Zur Einführung Θα ήθελα εισαγωγικά να αντιμετωπίσω τις ε, πιο πρόσφατες χρηματοπιστωτικές ε, εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Και στη συνέχεια θα είμαι διαθέσιμος να ασχοληθώ με τα θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν και εσάς συγκεκριμένα το, την εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση της κρίσης και επίσης τα θέματα των φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Έρχομαι τώρα σε μια γλώσσα που τη μιλάω λίγο καλύτερα. Μετά από την τελευταία μας ε, ακρόαση τον, Οκτώβριο με τον πρώην πρόεδρο Τρισέ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάρει μια σειρά μέτρων για να εξασφαλίσει ότι θα εξακολουθεί να εξασφαλίσει τη σταθερότητα τιμών σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο σε ένα περιβάλλον το οποίο παραμένει δύσκολο και προκλητικό. Τα μέτρα αυτά αφορούν αλλαγές τόσο στα επιτόκια όσο και στα λεγόμενα ατυπικά μέτρα, τα non-standard μέτρα για τα επιτόκια. Όπως ξέρετε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις αρχές Δεκεμβρίου αποφάσισε να μειώσει τα κύρια επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 25 σημεία βάσης. Μετά από μια αντίστοιχη μείωση πάλι κατά 25 σημεία βάση, δηλαδή 0,25% στις 3 Νοεμβρίου του 2011. Σε ό,τι αφορά την βραχυπρόθεσμη πορεία ανάπτυξης της περιοχής του ευρώ, οι μεγαλύτερε εντάσει που παρουσιάζονται στι χρηματαγορέ εξακολουθούν να τροχοπεδούν την οικονομική δραστηριότητα στον χώρο του ευρώ και οι προοπτικέ παραμένουν αβέβαιε. Η οικονομική δραστηριότητα τη περιοχή του ευρώ θα πρέπει να ανακάψει σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2012, όπως προβλέπεται και από το προσωπικό του ευρωσυστήματος, προσβλέφθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου. Εξακολουθούν όμως να παραμένουν πολλοί κίνδυνοι και κίνδυνοι να μην επιτευχθεί αυτή η ανάκαμψη για αυτή την προοπτική. Σε ό,τι αφορά τι εξελίξει των τιμών, ο πληθωρισμό ήταν 3% τον Νοέμβριο και προβλέπεται να παραμείνει πάνω από το 2% για τους επερχόμενου μήνες, πριν μειωθεί σε επίπεδα κάτω του 2% που είναι ακριβώς αυτό το οποίο προβλέπεται από τις αναλύσεις του ε, προσωπικού μας για το Δεκέμβριο, από το Δεκέμβριο λόγω αυτού του πλαισίου χαμηλότερης ανάπτυξης στην περιοχή του ευρώ και ε, των πιέσεων που υπάρχουν στα ημερομίσθια και τις τιμές θα πρέπει να παραμείνει περιορισμένος ο πληθωρισμός στην περιοχή του ευρώ. Οι κίνδυνοι για το μεσοπρόθεσμο διάστημα παραμένουν ισορροπημένοι. Τα τελευταία νομισματικά στοιχεία καταδεικνύουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές αν ξεπεράσουμε μονάχα το θέμα της βραχυπρόθεσμης διακύμανσης και ευμεταβλητότητος, η ανάλυση των νομισματικών θεμάτων δείχνει ότι θα παραμείνει περιορισμένη η ανάπτυξη της νομισματικής μάζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι αποφασισμένο να εξασφαλίσει ότι οι προσδοκίες σε σχέση με τον πληθωρισμό θα παραμείνουν μέσα στα πλαίσια του στόχου μας να διατηρήσουμε τον πληθωρισμό κάτω από αλλά πολύ κοντά στο 2% σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Έρχομαι τώρα σε ορισμένα μέτρα που πήραμε, τα ατυπικά μέτρα, τα μη στάνταρ μέτρα τα οποία ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να αναχαιτήσουν αρνητικές επιπτώσεις στο μηχανισμό μετάδοση τη νομισματική πολιτική που μπορεί να προκύπτουν από τι εντάσει σε ορισμένα τμήματα των χρηματαγορών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την πίεση που ασκείται στι χρηματαγορέ για την παροχή πιστώσεων στι επιχειρήσει και τα νοικοκυριά. Καταρχήν υπήρξαν μία σειρά από μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν για να εξασφαλίσουν ότι οι τράπεζες παραμένουν, ε, εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις χρηματαγορές. Αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε τριετής διαδικασίες αναχρηματοδότησης για να υποστηρίξουμε την παροχή πιστώσεων στην οικονομία της Ευρωπαϊκής της ζώνης του ευρώ. Τα μέτρα αυτά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ότι οι συνεχιζόμενες εντάσεις στις χρηματαγορές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα των τραπεζών στην περιοχή του ευρώ να εξασφαλίσουν αναχρηματοδότηση σε πιο μεγάλους χρονικούς ορίζοντες. Νωρίτερα τον Οκτώβριο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να έχουμε δύο πρόσθετες πράξεις ε, χρηματοδότησης με διάρκεια περίπου ένα έτος. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι σε όλες τις πράξεις αναχρηματοδότησης μέχρι τουλάχιστον το πρώτο μισό του 2012 όλη η ρευστότητα που θα το από τις τράπεζες θα εδίδεται πλήρως σε σταθερό επιτόκιο. Η χρηματοδότηση μέσω της αγοράς καλυπτωμένων ομολογίων επίσης διευκολύνεται από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Οκτώβριο να εισαχθεί ένα νέο σύστημα ένα νέο πρόγραμμα αγόραση καλυπτωμένων ομολογιών ύψου 40 δισεκατομμύριων ευρώ. Τέλος, η χρηματοδότηση σε αμερικανικά δολάρια διευκολύνεται με τη μείωση της, ε, ε, του τιμήματο των προσωρινών ε, συμφωνιών ανταλλαγής swap μεταξύ δολαρίων και ευρώ. Όλα αυτά τα πέντε μέτρα θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε σταθερή χρηματοδότηση και σε σε χρηματοδότηση μεγαλύτερης διάρκεια κάτι το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν να δανειοδοτούν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Το υπογραμμίζω αυτό. Να συνεχίσουν να υπογραμμίζουν και στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Δεύτερον, η πρόσβαση σε πράξεις αναχρηματοδότησης μπορεί για ορισμένε τράπεζες να περιορίζεται από την έλλειψη επαρκών εγγυήσεων. Για να ξεπεράσουμε το θέμα αυτό, έχει αποφασιστεί μια προσωρινή επέκταση του καταλόγου των επιλεξίμων εγγύησεων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει σαν στόχο να ενισχύσει τη χρήση των τραπεζικών διατραπεζικών δανείων ως εγγυήσει σε πράξεις του, Ευρωπα... του ευρωσυστήματος, του συστήματος του ευρώ. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να υποστηρίξουν τι δανειοδοτήσεις των τραπεζών, αυξάνοντα τον αριθμό το νόγκο μάλλον των στοιχείων ενεργητικού στα, ε, στους ισολογισμούς των τραπεζών που μπορούν να υποστηριχθούν και να χρησιμοποιηθούν ως εγκυοδοτήσεις για ε, δανεισμό από την Κεντρική Τράπεζα. Τρίτον, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενισχύσει την δράση των χρηματαγορών. Καταρχήν, το αποθεματικό, το λόγος αποθεματικού θα μειωθεί προσωρινά από το 2% στο 1%. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν περισσότερα κίνητρα για αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στην αγορά να συμμετάσχουν σε συναλλαγές των χρηματαγορών και αυξάνει συγχρόνως και την, ε, τις οι οποίες είναι διαθέσιμες για τις τράπεζες γιατί μειώνει τις ανάγκες χρηματοδότησής τους έναντι του ευρωσυστήματος και επομένως το επίπεδο ε, εγγυήσεων που θα πρέπει να ε, καλύπτει αυτές τις πράξεις δανειοδότηση από την Κυρική Τράπεζα. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν σαν στόχο να ενισχύσουν την πρόσβαση του τραπεζικού τομέα σε μεγαλύτερη ρευστότητα και να ευνοήσουν τη λειτουργία των χρηματαγορών στο, στη ζώνη του ευρώ και με τον τρόπο αυτό να περιορίσουν τους κινδύνους για την πραγματική οικονομία από την έλλειψη δυνατοτήτων χρηματοδότηση. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ότι τα επίσημα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα διαβιβαστούν πλήρως στην οικονομία, στη γενική οικονομία. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο και η σταθερότητα των τιμών. Έρχομαι τώρα στα συμπεράσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ήταν μια πραγματική τομή σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να παραμείνουμε δεσμευμένοι σε υγιείς και διαφανείς κανόνες για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν τεθεί τα θεμέλια ενός δημοσιονομικού συμβολέου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο είχε προταθεί και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν έγινε η ακρόαση της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας, στις Κεντρικής Τράπεζας στην αρχή αυτού του μήνα. Αποφασίστηκε το διαφθοντικό έλλειμμα των κρατών μερών να μην ξεπερνάει το 0,5% του ονομαστικού του ΑΕΠ οι χώρε τη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να εφαρμόσουν ένα κανόνα στο εθνικό τους νομικό πλαίσιο σε θεσμικό επίπεδο. Ο στόχο είναι να αποφευθούν υπερβολικά ελλείμματα πριν δημιουργηθούν και όχι να προσπαθεί κανείς να τα τυθασεύσει όταν έχουν αναδυθεί. Προβλέπεται επίση ένα αυτόματος διορθωτικός μηχανισμός εάν υπάρχουν υπερβάσεις αυτού του ορίου. Αποφάσισαν επίσης οι ηγέτες των κρατών και κυβερνήσεων να υπάρχει και ένα αριθμητικό ένας αριθμητικός γνώμονας για τη μείωση σε αιτήσιο επίπεδο του χρέους για να μειωθεί το επίπεδό του. Θα υπάρχουν αυτόματες κυρώσεις για τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ εάν ξεπενιέται το επίπεδο 3% για τα ελλείμματα. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να ζητηθεί από αυτό να ερμηνεύσει και να ελέγξει την εφαρμογή αυτών των κανόνων σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το νέο δημοσιονομικό συμβόλαιο είναι ένα σημαντικό μήνυμα γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια σαφή στροχιά για τη μελλοντική εξέλιξη της περιοχής του ευρώ. Αντιμετωπίζει τις προσδοκίες και των πολιτών και των χρηματαγορών. Το να έχουμε σαφείς κανόνες σε πρωτογενή νομοθεσία των κρατών μελών και να γίνονται εκτελεστοί και εφαρμοστεί, αυτοί οι κανόνες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όλα αυτά συμβάλλουν στο να γίνουν τα δημόσια οικονομικά των χωρών της του ευρώ πιο ανθεκτικά και ισχυρά. Αυτό το χαιρετίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε ό,τι αφορά τα εργαλεία για τη διαχείριση της κρίσης στη ζώνη του ευρώ, χαιρετίζουμε την απόφαση των κρατών των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ να ενισχυθεί ο μηχανισμός χρηματοοικονομικής σταθερότητας και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σε μια σειρά περιοχών. Πρώτον, υπάρχει τώρα μεγαλύτερη ευελιξία στη ζώνη του ευρώ για να μπορέσει να αναχαιτήσει τα προβλήματα γιατί θα εφαρμοστεί, σε, ε, θα εφαρμοστεί από τον Ιούλιο του 2012 το ESM, ο Ευρωπαϊκός Μηχανικός Σταθερότητος και όχι το 2013 όπως προβλεπόταν. Επίσης για το Ευρωπαϊκό ε, Μέσο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, το EFSF, θα παραμείνει ενεργό για όλα τα προγράμματα τα οποία είναι εν εξελίξη μέχρι τον Ιούλιο του 2013. Δεύτερον, Έχουμε μια διευκρίνηση <clears throat> ότι σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ιδιωτών πιστωτών, η Ευρωπαϊκή Ζώνη, <clears throat> ζώνη του ευρώ θα παραμείνει πιστή στις πρακτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κάτι το οποίο καθησυχάζει τους επενδυτές. Τρίτον, υπάρχει απόφαση να υπάρξει μια έκτακτη διαδικασία στους κανόνες ψηφοφορια του Ευρωπαϊκού ε, Μηχανισμού Σταθερότητας, παρά το γεγονο ότι υπόκειται ακόμα σε έγκριση από το Φιλανδικό Κοινοβούλιο. Και αυτό είναι σημαντικό για να είναι αποτελεσματική η λήψη αποφάσεων ιδίως σε καταστάσεις κρίσεων. Για το Ευρωπαϊκό Μέσο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε ότι η Κεντρική Τράπεζα θα είναι σε θέση να λειτουργεί ως πράκτορ του συστήματος αυτού στις ε, συναλλαγές στις χρηματαγορές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την υποστήριξη κατά πάσα πιθανότητα ενό αριθμού εθνικών κεντρικών τραπεζών θα δώσει την τεχνική τη υποδομή και την τεχνογνωσία τη στο EFSF, στο σύστημα χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Έχουν ήδη ξεκινήσει τεχνικέ και νομικέ προετοιμασίε για κάτι τέτοιο και ελπίζουμε μέχρι το τέλο του Ιανουαρίου να έχουν περατωθεί. Και έρχομαι εν τέλει στο τελευταίο θέμα που είναι οι φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι δραστηριότητες των φορέων αυτών, ιδίως σε ό,τι αφορά το, το κρατικό χρέος και το Ευρωπαϊκό Μέσο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχουν βρεθεί στο προσκήνιο πρόσφατα στην Ευρώπη. Υπήρξαν εκκλήσεις για καλύτερη ρύθμιση των φορέων αυτών. Με το, μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν για τους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκονται σε συζήτηση και στη δική σας Επιτροπή. Οι αξιολογήσεις έχουν μεγάλη επίπτωση στη λειτουργία της αγοράς και την ευρύτερη οικονομία. Το να υπάρχει ένα ανθεκτικό και υγιές πλαίσιο η αξιολόγηση είναι απαραίτητο. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να έχει σαν στόχο να εξυπηρετήσει τους εξής στόχους. Να μειώσει την υπερβολική διακύμανση στις αγορές, να βελτιώσει την ποιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης και τρίτον να επαναφέρει την εμπιστοσύνη των αγορών. Τα δύο θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά είναι πρώτον είναι καταρχήν το να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει η κατάλληλη βασική μεθοδολογία για την αξιολόγηση και επίσης ότι υπάρχει διαφάνεια των αξιολογήσεων. Και δεύτερον, το να μειώσουμε την μηχανιστική χρησιμοποίηση στην νομοθεσία και στις πρακτικές αγορές των αξιολογήσεων. Οι αξιολογήσεις είναι απλώς ένας τυφλοσούρτης που απλοποιεί πολλαπλές αξιολογήσεις κινδύνου. Αλλά θα πρέπει να είναι μόνο ένα από πολλά εργαλεία που θα έχουν οι επενδυτές. Δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα ε, χρηματοπιστωτικά, την ανάγκη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επενδυτές να κάνουν δικές τους αξιολογήσεις. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα αποφύγουμε μια μηχανιστική εξάρτηση από εξωτερικούς φορείς πιστολογικής αξιολόγησης. Τέλος, θα ήθελα να σας πω πώς χρησιμοποιούμε εμείς την Κεντρική Τράπεζα της Αξιολογήσης. Στην πράξη, για τα περισσότερα αξιόγραφα τα οποία βρισκόνται στην αγορά, όπως είναι παραδείγματος χάρη κρατικά ομόλογα, το πλαίσιο αξιολόγησης ε, ε πιστοληπτική ικανότητας χρησιμοποιεί κυρίως τις αξιολογήσεις επιλέξιμων φορέων αξιολόγησης, χωρίς όμως μηχανιστικά να βασίζεται σε αυτές τις αξιολογήσεις, διότι γνωρίζει τις μεθοδολογικές, τα μεθοδολογικά όρια αυτών των αξιολογήσεων. Επιφυλασσόμεθα πάντα τη δυνατότητα να απορρίψουμε ή να περιορίσουμε τη χρήση ορισμένων στοιχείων ενεργητικού επί τη βάση οποιασδήποτε πληροφορία σε σχέση με την πιστοληπτική αξία του, που μπορεί να έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε εφαρμόσει λοιπόν αυτή τη διακριτική ευχέρεια για να αναστείλουμε προσωπικά, προσωρινά, την ε, ανάγκη να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο αξιολόγηση για τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται ως ε, εγκυοδοσίες μετά από τη διαδικασία που έχει γίνει με προγράμματα προσαρμογής για ορισμένες κυβερνήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Uh, uh, ευχαριστώ. Έχω περισσότερες ερωτήσεις ε, από ότι διαθέσιμο χρόνο. Παρακαλώ, είστε σύντομοι. Έχουμε πεντά λεπτά. Θα διακόπτω με τα πέντα λεπτά. Ένα λεπτό για κάθε ερώτηση και τέσσερα λεπτά για απαντήσεις. Ακόμα και έτσι χρειαζόμαστε 110 λεπτά που δεν έχουμε. Πρώτο ερώτημα. Ο Ζων Πολ θέτει το πρώτο ερώτημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε για αυτό τον πρώτο νομισματικό, σε αυτό τον πρώτο νομισματικό διάλογο εξ ονόματος του ΕΛΚ. Και διαπιστώνουμε ότι οι εφημερίδες ήξεραν πριν από μας τι θα λέγατε. Θα ζητήσω λοιπόν το εξής. Να εκτιμήσετε τον τίτλο της εφημερίδας γιατί ο αρχισυντάκτης συνήθως γράφει τον τίτλο για να τραβήξει περισσότερο κόσμο. Ιδού λοιπόν ποιος είναι ο τίτλος του Financial Times σήμερα. Και από τις πρώτες γραμμές του άρθρου λέει ότι ενώ ο προκάτοχός σας έλεγε ότι είναι παράλογο αυτό το σενάριο, εσείς λέτε ότι πρέπει να μελετηθεί. Και γράφει η εφημερίδα λοιπόν αυτό που διαβάσατε κι εσείς, δώστε μου μερικές εξηγήσεις, πώς το ήξερε. Το ανέμενα αυτό το ερώτημα, το περίμενα. Έχετε δίκιο που τονίζετε, που δίνετε σημασία σε αυτό τον τίτλο. Όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, εκείνοι γράψανε τον τίτλο, όχι εγώ. Αλλά δεν αφιβάλλουν καθόλου, τουλάχιστον για την ισχύ του ευρώ, για την βιωσιμότητά του και για το ότι δεν μπορεί να καταργηθεί. Αυτό το έλεγε ήδη η συνθήκη του Μάστριχτ, ότι το ενιαίο νόμισμα δεν πισωγυρίζεται. Πολλοί όμως, ιδιαίτερα εκτός της Ευρωζώνης, ξοδεύουν πολύ χρόνο κάνοντας απλώς μάταιες σκέψεις, δηλαδή τι θα γινόταν αν, τι θα γινόταν αν, με καταστροφικά σενάρια για την Ευρωζώνη όλοι τους. Αντί να πούμε λοιπόν όχι, όχι δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει διατάραξη, εμείς λέμε γιατί. Πολλοί όμως το σκέφτονται. Μία ανάλυση του εξαιρετικά μεγάλου κόστους που θα σήμαινε μία ανατροπή είναι κάτι που το καταλαβαίνει ο καθένας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Ούντο τώρα. Καλώ ήρθατε κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θέλω να σα καλωσορίσω στην Επιτροπή μα. Θα ήθελα να σα θέσω ένα ερώτημα για του φορεί πιστοληπτική αξιολόγηση. Έχουν κρατήσει μια επικριτική στάση για πολλά κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και με την, ε, μετά την διάσκεψη τη 9η Δεκεμβρίου. Ακόμα και με την ε, Μεγάλη Βρετανία, αν αυτό δυνατό πολλοί συνάδελφοι όπως ο κύριος Ντομένης έχουν ζητήσει να υπάρξει στεναρή νομοθετική ρύθμιση για, αυτές τις, ε, για αυτές τις εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης. Αυτές οι εταιρείες θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να βγει από την κρίση. Ίσως θεωρούν ότι δεν υπάρχει μια επαρκής πολιτική θέληση και επαρκή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι θέλετε να πείτε λοιπόν για όλα αυτά και τι θα πείτε και στις, ε, σε όλους αυτούς που θέλουν ε, στην ε, Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα να πάρουν πιο φτηνές πιστώσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μπορούν να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη. Με ποιο τρόπο λοιπόν μπορεί να υποστηριχθεί από την Κεντρική Τράπεζα η διαδικασία ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτήσατε δύο πράγματα. Το ένα αφορά τους οίκους αξιολόγησης μπορεί κανείς να σχολιάσει ποικιλοτρόπως την ποιότητα και το χρονισμό των αξιολογήσεων αυτών. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε θετικά τις εμπειρίες που είχαμε με τους οίκους αξιολόγησης, κυρίως πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τούτων λεχθέντων πρέπει να διερωτηθούμε το σημαντικότερο ερώτημα που να θέσουμε. Πώ θα πηγαίναμε, πώ θα προχωρούσαμε χωρί αυτέ τι αξιολογήσει, τι θα έπρεπε να κάνουμε για να αντικαταστήσουμε τι αξιολογήσει των οίκων αξιολόγηση. Διότι θέλουμε να έχουμε πληρέστερο σύστημα αξιολογήσεω πιστοληπτικής πιστοληπτική ικανότητα αντί του συστήματο που έχουμε τώρα που βασιζόμαστε μόνο αξιολογήσει των φορέων αξιολόγηση. Το ερώτημα είναι, τι συγκεκριμένα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τους οίκους αξιολόγησης. Πρώτο βήμα είναι αυτό που θα κάνουν οι ρυθμιστικοί φορείς. Οι ρυθμιστικοί φορείς θα έπρεπε να μειώσουν την εξάρτηση των ρυθμίσεων από την αξιολόγηση των οίκων αξιολόγησης. Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό. Επί του παρόντος μπορεί να δει κανείς ότι η ρύθμιση ε, είναι ενταγμένη στις ε, ε αξιολογήσει των οίκων αξιολόγησης. Αν αλλάξουν οι αξιολογήσεις, έτσι αλλάζει και η ρύθμιση αυτομάτως των ρυθμιστικών φορέων. Νομίζω ότι αυτός ο αυτοματισμός θα πρέπει να μειωθεί. Θα έπρεπε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις αξιολογήσει των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγηση ε, σαν η μία από τις ροές ε, πληροφοριών, όχι μοναδική πληροφορία. Αυτό ισχύει για τους μυστικούς φορείς, αλλά ισχύει ακόμα περισσότερο αυτό για τους επενδυτές. Μπορούμε να δράσουμε όσον αφορά τους ρυθμιστικούς φορείς. Έχουμε ετοιμάσει διάφορα σχέδια με αυτό το στόχο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε εδώ και δύο χρόνια περίπου ο τίτλος ήταν πώς θα απαλλαχθούμε από τις αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης. Για τους επενδυτές δεν αρκεί να απαλλαγούμε από τις αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγηση, αλλά θα πρέπει να είναι κανείς ικανός να κάνει δική του εσωτερική, τη δική του αξιολόγηση. Ζητάμε από τις τράπεζες να το κάνουν επεκτείνουμε την χρήση των εσωτερικών συστημάτων αξιολόγησης. Το άλλο ερώτημα αφορούσε την ανάπτυξη. Και ανάπτυξη στις χώρες αυτές, τις συγκεκριμένες που αναφέρατε. Τα μέτρα που λάβαμε, πιστεύω, τις περασμένες εβδομάδες, πότε ήταν η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 8 του μηνός, Έχω σαν στόχο ακριβώς αυτό γνωρίζουμε ότι οι τράπεζες τώρα και εμείς περισσότερο στο μέλλον αντιμετωπίζουν περιορισμούς πάρα πολύ μεγάλους στον φάει χρηματοδότηση. Κυρίως το πρώτο τρίμηνο του 2012 αντιμετωπίσουν και όχι μόνο τότε. Όλος ο χρόνος θα είναι δύσκολος για τις τράπεζες. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε, πάση θυσία, είναι σοβαρή μείωση των πιστώσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περί περαιτέρω επιβράδυνση της ανάπτυξης και ενδεχόμενη ύφεση. Θέλουμε να το αποφύγουμε αυτό. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό. Αν μπορούμε όμως να μειώσουμε τις σηματοδοτικές πίεσεις, βρίσκουμε ένα σημαντικό ποσοστό της απάντησης που ζητάμε. Ευχαριστώ. Σιλβί Γκουλάρ, επόμενο ερώτημα. Bonjour, Monsieur le Président. Σάρων, εδώ είμαι. Καλώς ήρθατε στο, στο διάλογό μας. Εξ ονόματος της ομάδας φιλελευθέρων, ζητήσατε πράγματι στην Ολομέλεια τη νέα αυτή δημοσιονομική συμφωνία και ξέρετε ότι οι βουλευτές οι οποίοι ήταν εισηγητέ για τα έξι νομοθετήματα, για το ΕΞΠΑΚ, είχαν ήδη κάνει μια μάχη για να επιτύχουν αυτό το, αυτή την ιδέα. Το περιεχόμενο είναι πολύ σημαντικό όμως. Πώς θα εφαρμόσετε πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτό το περιεχόμενο με κάθε ανεξαρτησία για να καλύψετε δύο απαιτήσει. Πρώτα απ' όλα, τα μέτρα αυτά να είναι συνεκτικά και να έχουν νόημα σε οικονομικό επίπεδο και δεν είμαι σίγουρο ότι έχουν οικονομικό νόημα. Όπως είπατε, πλησιάζουμε σε μία ύφεση και αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις θα έχουν πόρους οι οποίοι μειώνονται. Δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη οι πρόοδοι που έγιναν για την μακροοικονομική εποπτεία Όλα αυτά λοιπόν έχουν χαθεί. Επανερχόμαστε σε μία πάρα πολύ στενή αντιμετώπιση της δημοσιονομικής λιτότητας. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πραγματικά ανεπαρκή. Το κείμενο που κυκλοφόρησε την, ε, την ε, Παρασκευή έχει σαφείς ελλείψεις. Ναι, Σάρων, συγγνώμη που μακρηγορώ. Υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των πάρα πολύ αυστηρών κριτηρίων και από του πάρα πολύ διάχυτου και ασαφούς μπλα μπλα και το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και από νομική έποψη. Και γι' αυτό ζητώ κύριε Πρόεδρε να σκεφτείτε και το θέμα της δημοκρατίας. Νομίζω ότι δεν μπορεί να προκύψει τίποτα το σταθερό και το μόνιμο στην Ευρώπη αν οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν πιστεύουν ότι οι αποφάσεις οι οποίες τους επιβάλλονται δεν έχουν τη σωστή δημόσια συζήτηση στο απαραίτητο επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστεί αυτό. Εγώ με μια απλή συγγήτρια μονάχα αλλά εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ζητήσω την κύρωση αυτού του κειμένου που πέρασε την προηγούμενη Παρασκευή. Οι ευρωπαϊστές δεν μπορούν να δεχτούν αυτή τη φάτσα. Και εσείς ήσασταν μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σταθερότητας. Καταλαβαίνει ένας Αμερικανός ή ένας Κινέζος τι αποφάσεις ελήφθησαν και τι σημαίνουν. Um, I, I think... Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το ερώτημά σα. Για να αντιμετωπίσω πρώτα την οικονομική ουσία του ερωτήματος που θέσατε και μετά θα περάσω στο πιο θεσμικό και πολιτικό περιεχόμενο του ερωτήματός σας. Δεν υπάρχει κάποια ισορροπία μεταξύ της λιτότητος και της ανάπτυξης. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη συνταγή που θα εξασφαλίσει και τα δύο. Η λιτότητα σημαίνει, μια βραχυπρόθεσμη οικονομική συρρήκνωση. Δεν μπορεί να το διαμφισβητήσει κανείς αυτό. Αλλά πρέπει να θέσουμε το ερώτημα. Είναι αυτό κάτι το οποίο μπορούμε να το αποφύγουμε ή όχι. Ήταν βιώσιμη η προηγούμενη κατάσταση. Λοιπόν, δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία επιλογή. Ότι θα προκαλέσει μια συρρήκνωση η λιτότητα, αυτό είναι σαφές. Στη συνέχεια, τι θα πρέπει να κάνουμε για να μετριάσουμε αυτή τη συρρήκνωση και τελικά να την αντισταθμίσουμε και να την ανατρέψουμε. Εδώ υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Καταρχήν, αν η κατάσταση του προϋπολογισμού σε μια χώρα είναι, αν η δημοσιονομική κατάσταση δεν είναι βιώσιμη, βλέπετε ότι η συρρήκνωση αυτή που έρχεται από την αύξηση των spread στο δημόσιο χρέος γίνεται πάρα πολύ ψηλή. Επομένω, η πρώτη κίνηση πρέπει να γίνει από τι εθνικέ κυβερνήσει και πολλέ εθνικέ κυβερνήσει δρούν και με το σωστό τρόπο και εμεί έχουμε χαιρετήσει τι εξελίξει οι οποίε έχουν γίνει σε κάποιε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να βλέπετε και την αρχή της ε, δημιουργίας μιας εμπιστοσύνης, όπου οι αγορές και οι άλλες χώρες αρχίζουν να νιώθουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από αυτές τις εξέλιξεις. Βλέπουμε βέβαια ότι δεν είναι αυτό γιατί χρειάζονται και δύο ακόμα στοιχεία τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν. Οι λιτότητα σε επίπεδο μιας χώρας και μόνο δεν πρόκειται να αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Θα πρέπει να υπάρξει πρόοδο στην οικονομική διακυβέρνηση όλης της Ένωσης, σαν δημοσιονομικής Ένωσης. Πρέπει να υπάρξει αυτό το λεγόμενο δημοσιονομικό συμβόλαιο. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα βασικό στοιχείο. Αν θέλετε να επανέλθει η εμπιστοσύνη των αγορών, πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη στη σύνολη ζώνη του ευρώ και μεταξύ των χωρών, μεταξύ πολιτών και κυβερνήσεων. Επίσης, για να επανέλθει αυτή η εμπιστοσύνη θα πρέπει να εφαρμοστεί ένας σωστός μηχανισμός, αυτό το δημοσιονομικό συμβόλαιο. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτό μονάχα σε σχέση με τα θέματα του προϋπολογισμού. Και αυτό ήταν το κομμάτι του six pack των έξι νομοθετημάτων που υλοποιήθηκε, που θα υλοποιηθεί καλύτερα σε νομοθετικό επίπεδο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι υπάρχει και ένα δεύτερο τμήμα, που είναι το μακροοικονομικό κομμάτι. Δεν θα πρέπει να το παραγνωρίσουμε. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μεταφράσουμε και το μακροοικονομικό κομμάτι σε πρωτογενή νομοθεσία. Αυτό δεν είναι εύκολο από ενοιολογική έποψη είναι ακόμα πιο δύσκολο από ότι η λιτότητα του προπολογισμού να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ τονίζω πάντα την ανάγκη να έχουμε μια παρόμοια αντιμετώπιση των μακροοικονομικών μεταρρυθμίσεων όπως κάνουμε και για τα θέματα λιτότητας. Αυτό το υποστηρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Δεν μπορώ λοιπόν παρά να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Αλλά όταν έχει κανείς και τις δύο αυτές ε, βάσεις θα πρέπει να έχουμε τις μεταρρυθμίσεις σε διαφθορτικό επίπεδο που θα αυξήσουν την οικονομική μεγένθηση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να θεσπίσουμε και ένα σύστημα σαν και αυτό που περιγράψετε πριν από λίγο. Αυτό θα βοηθήσει ιδίω τις θεσμικά φτωχές χώρες, οι, αυτές που έχουν θεσμικά προβλήματα, να αντιμετωπίσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις που από πολιτική έποψη είναι πάρα πολύ οδυνηρές και δύσκολες. Ευχαριστώ. Ήδη έχουμε καθυστερήσει 1,5 λεπτό, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε για τα θεσμικά όργανα. Θα απαντήσετε για την ανάγκη να έχουμε δημοκρατία. Σίγουρα. Δεν θα το αμφισβητήσω αυτό. Σίγουρα. Όχι, δεν το μόνο ECR Κύριε Ντράγκη, την περασμένη εβδομάδα, Φρανσουά Ρολάντ, ο ε, για την υποψήφια στην Ελληνική Προεδρία είπε ότι εάν εκλεγεί θα ήθελε να παροτρύνει να αγοράσει κρατικά ε, ομόλογα περισσότερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να χρησιμοποιήσει την ισχύ πυρό τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο κύριο Ρολάντ έγραψε ένα βιβλίο για να προωθήσει την υποψηφιότητά του. Το γαλλικό όνειρο είναι ο τίτλος. και χρειάζεται ένα βιβλίο για να καταλάβει κανείς το γαλλικό όνειρο. Είναι απλό. Είναι τελικά ε, το χρήμα. Θέλει να δώσετε τα χρήματα για το βούτυρο. Το, το, βούτυρο και το χρήμα του βουτύρου. Είναι η ώρα του, του Χριστουγέννου, τα Ι Βασίλη και δεν μου φαίνεται ότι είσαι Ι Βασίλης. Και θέλετε να, κύριε θέλετε να γίνετε ε, και κάτι τέτοιο. Να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Και αυτό που είπε λοιπόν, αυτό που αναφέρθηκε και την έκκληση που απευθύνω όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πώς τα βλέπετε. Κοιτάξτε, θέλω να υπενθυμίσω προς όλους ότι η συνθήκη προσδιορίζει πολύ συγκεκριμένα ποια είναι η εντολή μας, δηλαδή να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα. Επίσης απαγορεύει χρηματοδοτήσεις νομισματικές και όπως είδατε θέλουμε να σεβαστούμε τη συνθήκη. Οποιαδήποτε άλλα μέτρα θα ήταν παραβίαση της συνθήκης και θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία του θεσμού μας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Αν χαθεί η αξιοπιστία, ιδιαίτερα της Κεντρικής Τράπεζας, δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει καθόλου και την εμπιστοσύνη των αγορών ή γενικότερα τη λειτουργία της Ευρωζώνης. Ευχαριστούμε, Σφέν. Καλώς ήλθατε και από τους πράσινους κύριε Δράκη θέλω να σας χαιρετήσω Χαίρομαι για ένα πράγμα σήμερα, γιατί έχουμε διαπιστώσουμε, έχουμε διαπιστώσει ότι μιλάμε και σε αυτή την Επιτροπή γερμανικά. Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι η εξής. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι συγχρόνως σε πάρα πολύ σημαντικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης γίνεται πίεση για εξοικονόμηση, ενώ η μακροοικονομική εικόνα βρίσκεται σε, στάση, σε φάση κάμψης. Θέλουμε να υποβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο την μακροοικονομική κατάσταση με τέτοια μέτρα. Και ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το θέμα αυτό. Μετά από το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε πει ο κ. Σαρκοζή ότι είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει φθηνό χρήμα στα κράτη-μέλη με 1% αλλά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες να πληρώσουν επιτόκια <clears throat> της τάξης του 7% όπως έγινε και η περίπτωση της ε, Ιταλίας. Ποια είναι η αποψή σα για να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σαν τράπεζα το EFSF, το μέσο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, και αν αυτό θα μπορέσει να μειώσει την πίεση για την χρηματοδότηση των ε, κρατών μέσω μονάχα των τραπεζών. Κοιτάξτε, το είπα και πριν. Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι είναι συρρήκνωση η λιτότητα. Δεν χρειάζεται να το αμφισβητήσουμε αυτό. Θέλουμε όμως η συρρήκνωση αυτή να είναι βραχυπρόθεσμη, προσωρινή και θέλουμε να ενεργοποιήσουμε όλα τα εργαλεία και κανάλια που υπάρχουν που να καταλήξουν στην επιστροφή των αγορών σε εμπιστοσύνη, μείωση του κόστους των δανείων και τελικά δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης. Για να υπάρξουν όλα αυτά πρέπει να υπάρξει πρώτα η, αυστηρότητα, η λιτότητα, να υπάρξει έλεγχος των προϋπολογισμών. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει επίσης να υπάρχει ένα γενικότερο όραμα, πρόγραμμα για να διασφαλίσουμε στους πολίτες της Ευρώπης την επίτευξη αυτών των στόχων και για τις αγορές. Πρέπει γι' αυτό να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές. Διότι τα τελευταία δέκα χρόνια υπήρξαν χώρες όπου ήταν πολύ χαμηλά τα επιτόκια, σχεδόν μηδέν και δεν αναπτύχθηκαν. Ανέβηκαν τα επιτόκια, πάλι δεν αναπτύχθηκαν. Ξανακατέβηκαν, πάλι δεν αναπτύχθηκαν. Η ανάπτυξή τους ήταν μηδενική σχεδόν και κάτω από το μηδέν για 10 χρόνια. Σε αυτές του είδου τις χώρες το θέμα δεν είναι κυρίως τα επιτόκια. Τα επιτόκια μπορεί να παίξουν ένα ρόλο αργότερα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει το μπλοκάρισμα που δημιουργείται από προστατευμένα συμφέροντα, από έλλειψη ανταγωνιστικότητας και ανταγωνισμού, από αγορές εργασίας που δεν λειτουργούν και αυτό βέβαια βλάπτει κυρίως τους νέους. Βλέπετε ότι σε αυτού του είδους τις χώρες το να ΕΠ είναι χαμηλότερο τώρα σε σύγκριση με 10 χρόνια πριν. Τώρα οι νέοι ιδίω κερδίζουν λιγότερα από ό,τι κέρδιζαν πριν από 10 χρόνια ή και 15 χρόνια. Για αυτές λοιπόν τις χώρες πρέπει κυρίως να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές. Βέβαια η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Με τις αποφάσεις που μόλις ελήφθησαν προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε μια νέα κρίση των, της που να οφείλεται σε έλλειψη χρημάτων. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα γιατί υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορεί να εξηγούν μια τέτοια κρίση. Εμείς όμως μιλάμε εδώ για τη χρηματοδότηση που για μένα είναι το σημαντικότερο κριτήριο. Και από τα μέτρα που ελήφθησαν φαίνεται ότι αυτό θα δουλέψει. Τέλος, ο τρίτος για να το πω έτσι πυλώνας μετά από την εθνική πολιτική και τα προγράμματα ενωσιακού επίπεδου υπάρχει ανάγκη ενός προστατευτικού τείχου σαν firewall που με επαρκή μέτρα να καταπολεμήσει την προσωρινή αστάθεια στις χρηματαγορές. Και το τελευταίο, η τελευταία διάσκεψη ανέφερε πολλά στοιχεία προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρώτον επιβεβαίωσε ότι το ESM θα εφαρμοστεί νωρίτερα από ό,τι είχαμε πει πριν και ότι το EFSF πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί επαρκώς το Μάρτιο, σε τρεις μήνες από τώρα. Δεν μιλάει πια συμμετοχή για συμμετοχή ιδιωτών. Γιατί υπάρχει το κύριο πρόβλημα της ε, αξιοπιστίας των χωρών. Υπάρχει το έλλειμμα και Γενικά, τα μέτρα που πρόβλεψε, που, στα οποία κατέληξε η διάσκεψη δεν είναι αρνητικά. Εγώ όμως ρώτησα τι φρονείται για τις άδειες που δίνουν για το EFSF, ναι, για το EFSF e ναι. και τις τράπεζες. Όχι, δεν νομίζω ότι έτσι ούτε παραβιάζουμε και καλυμμένα ούτε φανερά τη συνθήκη η ΕΚΤ θέλει να διασφαλίσει την νομισματική σταθερότητα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει χωρίς να υπονομεύει, χωρίς να αποδυναμώνει την αξιοπιστία του θεσμού. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ο Νικόλας. Έλληνας είναι. Ράγκη, όπως ξέρετε, σύμφωνα με την απόφαση της 26ης του Οκτωβρίου, το χρέος της Ελλάδας που ανήκει στον ιδιωτικό τομέα θα κουρευτεί κατά 50%. Ταυτόχρονα υπάρχει απόφαση συμμετοχής του ιδιωτικού φορέα των ιδιωτών σε αυτό το κούρεμα, το λεγόμενο PSI, αναφερθήκατε πριν, και ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2012 για να ενεργοποιηθεί η Συμφωνία για τη Νέα Δανειακή Σύμβαση και Βοήθεια για την Ελλάδα. Από όσο ξέρουμε, η ελληνική κυβέρνηση σε αυτούς που αναφέρεται το κούρεμα τους προσφέρει ομόλογα που τα εγγυάται το EFSF. Αλλά το EFSF, όπως κουβεντιάζουμε, είναι στην κρίση και σε κίνδυνο υποβάθμισης, όπως αρκετές χώρες που μετέχουν σε αυτό το μηχανισμό και παρέχουν τις μεγαλύτερες εγγύησεις. Και το ερώτημα είναι τώρα, γιατί και ποιοι ομολογούχοι θα δέχονταν ένα τέτοιο κούρεμα απέναντι σε αμφίβολες εγγυήσεις και το δεύτερο ίσως πιο προσωπικό. Εσείς πώς θα τους πείθατε αυτούς τους ομολογιούχους να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να δεχτούν το κούρεμα και μάλιστα σε ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Well, I, I, I actually can't δεν μπορώ να κάνω πολλά σχόλια επ' αυτού, εφόσον οι συζητήσεις για το PSI ε, ε, λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή. Αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι μεταξύ της ελληνικής κυβερνήσεως και των τραπεζών. Αλλά μπορώ να σας πω ότι όσον αφορά το FSF, το FSF είναι έτοιμο να δράσει. Και το ότι τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιεί και θέτει στην διάθεση του FSF τις υποδομές της και την τεχνογνωσία της, αυτό είναι κάτι που κατά κάποιο τρόπο εξασφαλίζει ότι θα έρθει τη στιγμή το FSF είναι εκεί για να δώσει τους αναγκαίους πόρους. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ντράγκη που μας εξηγήσατε σήμερα την όλη κατάσταση. Στο Βερολίνο την περασμένη εβδομάδα είπατε ότι οι χώρες θα πρέπει να σώσουν τους εαυτούς τους. Δεν θα πρέπει να περιμένουν να βρουν έναν εξωτερικό σωτήρα. Αυτό πιστεύει το πολιτικό μου κόμμα, δηλαδή το κόμμα ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Πιστεύει ότι οι χώρες θα πρέπει να βοηθήσουν τους εαυτούς τους. Όμως επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο ελέγχει το δικό του νόμισμα και έχει τη δική του κεντρική τράπεζα, έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τη δική του νομισματική πολιτική. Αυτή η ελευθερία δεν υπάρχει για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Καλείται χώρες με υψηλή ανεργία να σωθούν, να σώσουν τους εαυτούς τους. Ταυτόχρονα όμως δεν χαλαρώνεται, δεν απελευθερώνεται την παροχή χρήματος. Λέτε ότι η λύση είναι η λιτότητα για τις χώρες. Δεν χρειάζεται μια εναλλακτική δίωδος να εγκαταλείψουν παραδείγματος χάρη την Ευρωζώνη, να υπονομεύσουν το εθνικό τους νόμισμα και να γίνουν εκ νέου ανταγωνιστικότερες οι χώρες και να ξαναδημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης για το λαό τους. Ευχαριστώ. Απάντηση. Είδα άλλη μια αναφορά στην συνέντευξη που έδωσα στο Financial Times. Όπως προανέφερα, δεν υπάρχει αντάλλαγμα μεταξύ λιτότητας και ανάπτυξης. Αν μειώσει μόνο τον προπολογισμό, αυξάνοντα του φόρου πιθανότατα και δεν κάνει τίποτα άλλο, σίγουρα δεν θα έχει όχι μόνο βραχυπρόθεσμη συρρήκνωση τη οικονομία, αλλά μεσοπρόθεσμη ύφεση. Α το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά αν κάνει κανείς όλες τις διαφορετικέ αλλαγές που χρειάζονται, αν αυτό που γίνεται σε εθνικό επίπεδο συνοδεύεται από πρόοδο σε, κο επίπεδο και όπως είπατε δεν αληθεύει η νομισματική μας πολιτική έγινε περιοριστική. Αντιθέτως μάλιστα είναι αρκετά χαλαρή και τα μέτρα που λάβαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου θα δείξει την ισχύ των μέτρων ξεκινώντας από αύριο. Πέραν αυτού Ακόμα και χωρίς να περιμένουμε για το μέλλον, η μείωση των επιτοκίων, η μείωση των, του ποσοστού αποθεματικών, η διεύρυνση των εγγυήσεων, ήδη, η αύξηση των εγγυήσεων ήδη υπάρχουν. Μη λησμονείτε από την άλλη ότι θα πρέπει να κινούμεθα εντός των ορίων των συνθήκων. Εντός των ορίων αυτών έχουμε παράσχει ε, μία ένα σημαντικό εργαλείο για την νομισματική πολιτική με τις αποφάσεις που ελήφθησαν που θα μπορούσε να βοηθήσει όλη την Ευρωζώνη αλλά και ιδιαίτερο στις χώρες που αντιμετωπίζουν την κατάσταση που περιγράψατε προηγουμένως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χωζέ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μία από τις πιο ωραίες ε, στα πιο ωραία μέρη τη Καζαμπλάνκας λένε «Αχ, τι ωραία που να ήμασταν στο Παρίσι». Βρισκόμαστε σε μια φάση που θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα του χρέου γιατί κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε συρρήκνωση των πιστώσεων και σε γενική ύφεση. Αυτό το οποίο μας μένει αυτή τη στιγμή είναι μονάχα η Κεντρική Τράπεζα. Το Ταμείο Σταθερότητος και Έκτακτης Επέμβασης Κανεί δεν ξέρει πότε θα λειτουργήσει, πώ θα λειτουργήσει. Ακόμα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα σταθερότητα δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει και αυτό να λειτουργήσει πλήρω. Η Κεντρική Τράπεζα αγοράζει κρατικό χρέο, Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι πού μπορεί να συνεχίσει να αγοράζει χρέος για έκτακτε λόγω έκτακτη ανάγκη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αγορές από την Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι το πρόβλημα αν αγοράζουμε ή όχι. Το θέμα είναι ποιο είναι το όριο. Να σας δώσω την εξής απάντηση. Γιατί έχουμε καταρχήν δώσει τόση σημασία στα θέματα των τραπεζών. Οι τράπεζες είναι περίπου 80% των δανειοδοτήσεων στην ζώνη του ευρώ. Είναι διαφορετικά τα πράγματα από ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου οι επιχειρήσεις και τα νοικοχειριά δανείζονται πολύ περισσότερο από τις, κεφα... από τις χρηματαγορές και όχι από τις τράπεζες. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι στον χώρο της Ευρώπης οι τράπεζες είναι σημαντικές για την πιστοδότηση. Επίσης, πρέπει να πω το εξή. Όταν βλέπει κανεί τι τράπεζες, βλέπει κανεί ότι οι μικρότερες και οι μεσαίε τράπεζες είναι, είναι αυτές οι οποίες έχουν εστιάσει τη χρηματοδότησή τους στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Επομένως, για να έχουμε τη δυνατότητα, για να βοηθήσουμε το τραπεζικό σύστημα να ξεπεράσει τις πιέσεις χρηματοδότησης, είναι σημαντικό γιατί θα βοηθήσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες εξαρτώνται από τις μικρομεσαίες τράπεζες. Αυτό είναι και ο στόχος των μέτρων τα οποία λάβαμε. Το επόμενο ερώτημα είναι το εξής. Ας υποθέσουμε ότι επιτυγχάνουμε τι θα κάνουν οι τράπεζες με τα χρήματα τα οποία παίρνουν. Όπως είπα πολλές φορές, ο πρώτος στόχος μας είναι να βοηθήσουμε να επανέλθει η χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί εκεί χρειάστηκε να εργαστούμε σκληρά για να αποφύγουμε μια ακόμα μεγαλύτερη σύρρυκνωση της ανάπτυξης από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Μπορούν οι τράπεζες να επαναγοράσουν τα ομόλογα που έχουν εκδώσει αυτά ή μπορούν να ε, αγοράσουν ομόλογα τα οποία καλύπτονται από κάποιες εγγύησεις. Το βασικό είναι ότι πρέπει οι τράπεζες να αποφασίσουν οι ίδιες ποια είναι η καλύτερη δράση τους στις επενδύσεις και στη δανειοδότησή τους ακολουθώντας το δικό τους μοντέλο επιχειρήσεων, την κερδοφορία τους, τις στρατηγικές της κτλ. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουν. Δεν ξέρουμε πόσα ομόλογα θα επαναγοράσουν λοιπόν οι τράπεζες. Το ερώτημά μου ήταν η Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα δεν αγοράζει ομόλογα με αυτό το διάβλο. Νο, συγγνώμη, πρέπει να παραξήγησα το ερώτημά σας. Μιλήσατε για τις αγορές στην δευτερογενή αγορά. Αλλά αυτές οι αγορές έχουν γίνει για να εξασφαλιστεί η επαναφορά της σταθερότητας, αυτό ήταν ένα προσωρινό μέτρο, δεν είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει το διενεκές. Όταν λέτε για το αν υπάρχει ένα όριο, φυσικά. Δεν έχει τεθεί κάποιο όριο, αλλά δεν έχει πει κανείς ότι αυτές οι αγορές θα είναι μόνιμες. Δεν είναι ούτε αιώνιες, ούτε χωρίς ποσοτικό όριο αυτές οι αγορές. Συγγνώμη γιατί δεν κατάλαβα καλά το ερώτημά σας. Ο Αντολίν Σάντσες Περσέδο, Ευχαριστώ και εγώ θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να χαιρετήσω τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας με την ευκαιρία της πρώτης παρουσίας του εδώ στο νομισματικό διάλογο και σας εύχομαι και καλές διακοπές, χριστιαγεννιάτικες διακοπές. Αυτό ισχύει για όλους τους Ευρωπαίους. Θα είναι πολύ θετικό να μπορούν να είναι καλές διακοπές. οι πληροφορίες που έχω, αυτή τη στιγμή έχετε κίνδυνους στο χαρτοφυλάκιό σας που είναι πολύ χαμηλότεροι από αυτούς που έχει η Federal Reserve στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλική Κεντρική Τράπεζα ή η Τράπεζα της Ιαπωνίας. Είναι σωστό αυτό. Και εάν υπάρχουν ακόμα εντάσεις στην αγορά είναι γιατί οι φορείς αξιολόγησης και οι αγορές δεν εκτιμούν την λευστότητα που δίνεται στις τράπεζες. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποια είναι η δική σας άποψη για το σημείο αυτό. Και τέλος, το πρόβλημα της νομισματικής πολιτικής είναι ότι στις καλές χρονικές στιγμές τα πράγματα είναι πολύ καλά για τις κεντρικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες δεν είναι τόσο κεντρικές και επομένως τα χαμηλά επιτόκια οδηγούν σε φούσκες που τελικά όλα αυτά τους οδηγούν στο να πληρώνουν αυτή τη στιγμή, στις δύσκολες στιγμές να πληρώνουν υψηλότερα επιτόκια. Υπάρχει κάποιος τρόπος να αναχαιτήσετε αυτή την ε, υπερκυκλική συμπεριφορά στην ε, ζώνη του ευρώ. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας για τα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ και ανταποδίδω και σε εσά και σε όλους τους υπόλοιπους. Να προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημά σας. Όσον αφορά τι αποφάσει που λάβαμε την περασμένη εβδομάδα για την νομισματική πολιτική, ποιο ήταν, ποιος ήταν ο στόχο. Θέλαμε να αντιμετωπίσουμε τι χρηματοδοτικέ πιέσει και του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης και την μείωση των πιστώσεων. Για να σας δώσω μια ιδέα για την πίεση. Έχουμε 230 δις ευρώ ομολόγων τραπεζικών μόνο το πρώτο, θα χρησιμοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους και περίπου 250-300 που θα πρέπει να εξοφληθούν στις αρχές του επόμενου έτους, το συγγνώμη. Και μετά έχουμε περίπου 200 συν δις ευρώ των CLOs που είναι αξιόγραφα εγγύσεων που εκδίδονται από επιχειρήσει που εκδίδονται και έχουν να πληρωθούν κατά τη διάρκεια του έτους, όχι το πρώτο τρίμηνο. Η αγορά ομολόγων λοιπόν θα έχει τεράστιες πίεσεις. Ανευπροηγουμένου ενδεχομένως. Στόχος μας, ποιος είναι, έχουν και άλλες, άλλα προβλήματα οι τράπεζες. Προέρχονται από έλλειψη κεφαλαίων τα προβλήματα τα άλλα είχαμε εντοπίσει κεφαλοχικές ανάγκες ε, των τραπεζών που υπήρχαν. Και από πλευράς κεφαλαίου τι θα μπουν σε πειρασμό να πουν οι τράπεζες. Είναι πολύ δύσκολο να μαζέψουμε κεφάλαια από τις αγορές σε αυτές τις τιμέ. Μπορώ να πουλήσω κάποια στοιχεία ενεργητικού. Καταρχήν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αλλά ο κίνδυνος να κάνει κανείς ξεπούλημα, όπω αποκαλείται, δηλαδή πωλήσει σε πολύ χαμηλές τιμές που θα δημιουργούσαν αυτές κατοφερική πορεία των τιμών θα ήταν ενδεχόμενο. Και το τρίτο κακό ενδεχόμενο, να μειώσουν τη δανειοδότηση τράπεζε απλούστατα. Μείωση δανειοδότησης. Και πέρα των πιέσεων από τα κεφάλαια, έχουμε και πιέσει από τη χρηματοδότηση. Τα μέτρα που πήραμε α, στις 8 Δεκεμβρίου ανταποκρίνονται στο δεύτερο τμήμα. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον η χρηματοδότηση των τραπεζών ε, καλύπτεται το πρόβλημα της χρηματοδότησης των τραπεζών κατά κάποιο τρόπο. Και υπάρχει και άλλη όψη. Όσον αφορά τα, ένα από τα προβλήματα που βλέπουμε τα εμπόδια ε, όσον αφορά τις πιστώσεις σήμερα εξαρτάται από την προσπάθεια αποφυγής ψηλού κινδύνου δεν εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον και αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη δεν δανείζει ο ένας τον άλλον. Οι τράπεζες δεν δανείζουν σε τράπεζες, δανείζουν σε πολίτες και δεν δανείζουν οι τράπεζες σε εταιρείε. Κάποιο από αυτό το πρόβλημα, από αυτή την αποφυγή ψηλού κινδύνου εξαρτάται στο ότι τράπεζα, μια τράπεζα θεωρεί ότι άλλη τράπεζα δεν έχει χρήματα. Ανησυχεί λοιπόν για τη ρευστότητα και αυτό μπορεί να μεταμορφωθεί σε ανησυχία όσον αφορά τη φερεγκαιότητα. Και τα μέτρα που πήραμε στις 8 Δεκεμβρίου καλύπτουν και αυτή την πτυχή του τραπεζικού συστήματος. Αυτή είναι η βασική λόγη. Ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο ε, θα αποφύγουμε κάποια μεγάλη κρίση πιστοτική, κάποιο πιστοτικό γεγονός. Εντάξει, ευχαριστώ. Α, Κάποιο άλλο τμήμα έχετε το ερώτημά σας, κάποια άλλη πτυχή. Αν οι αγορές αξιολογούν σωστά το επίπεδο του κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντηση, δύσκολο να το πούμε αυτό. Ούτε ναι, ούτε όχι είναι η απάντηση. Να σας πω ποιο είναι το ιστορικό των προσφάτων γεγονότων. Επί σειρά ετών, τα επιτόκια της αγοράς δεν αντικατόπτριζαν τις διαφορές μεταξύ χωρών. Είχαμε χώρες. Όταν δημιουργήθηκε το ευρώ, είχαμε χώρες με, που, ε, στις οποίες επικρατούσαν πολύ ε, διαφορετικές αρχικές συνθήκες. Είχαμε χώρες με, πολύ, με τεράστιο χρέος και άλλες με μικρό χρέος. Χώρες με μεγάλη ανάπτυξη και χώρες χωρίς ανάπτυξη. Και οι πολιτικές επίκυλαν. Σε κάποιες χώρες οι πολιτικές ήταν λίγο πολύ συγκράτηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα, αύξηση παραγωγικότητας. Σε άλλες χώρες η πολιτική ήταν α, έλλειψη ελέγχου των προπολογισμών. Παρ' όλα αυτά τα επιτόκια δεν αντικατόπτυζαν τις διαφορές κινδύνων που υπήρχαν. Άρα τελικά υποτίμησαν τη διαφορά των κινδύνων. Μετά είχαμε την κρίση των Lehman Brothers, την κρίση του 2007-2010 και εκεί άλλαξε εντελώς η αντίληψη από πλευρά επενδυτών και αγορών του κινδύνου. Κατάλαβαν ξαφνικά την μεγάλη υποτίμηση του, του, του κινδύνου σε διάφορες χώρες. Και τώρα υπερβάλλουν όσον αφορά την αποτίμηση του κινδύνου. Είναι μια άποψη που εξέφρασα επανειλημμένα Δηλαδή, οι τώρα ε, τιμές των κρατικών ομολόγων αντικατοπτρίζουν μια κρίση. Δεν θα ήταν οι τιμές που θα βλέπαμε σε κανονικές εποχές. Όμως, ε, δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στις ε, πρώτερες συνθήκες. Θα πρέπει να μάθουμε ότι υπάρχουν spreads και ότι τα spreads θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον κίνδυνο και το πώς λειτουργούν τα spreads στην αγορά είναι κάτι υγιές, διότι στέλνουν μήνυμα σε εκεί που μορφώνουν την πολιτική σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι δείχνουν ότι πρέπει να επιταχύνουν την πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Ραμόν, παρακαλώ να περιοριστείτε σε μία ερώτηση. Οι οι συνάδελφοι που ακολουθούν τον κατάλογο θα χάσουν τη θέση του. Ευχαριστώ πολύ. Από το Μάιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει κρατικά ομόλογα των κρατών μελών στις αγορές. Εγώ υποστηρίζω απόλυτα αυτή την παρέμβαση και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τον τρόπο αυτό έχει σώσει το ευρώ. Αλλά υπάρχουν κάποιες χώρες στις οποίες αυτές οι παρεμβάσεις μπορεί να έχουν δημιουργήσει κίνητρα για να καθυστερήσουν οι διαρθωτικές αλλαγές. Έρχομαι από τη Βαρκελόνη, κύριε και η κυβέρνηση της ε, Καταλωνίας έχει θέσει σε ισχύ ένα πρόγραμμα προσαρμογής που έχει μειώσει κατά 10% τις δαπάνες και του χρόνου θα τις μειώσει κατά περαιτέρω 5% για να επιτύχει το στόχο ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Αλλά η κυβέρνηση Καταλωνίας έχει να αντιμετωπίσει σήμερα προβλήματα ρευστότητας γιατί μειώνται οι μεταφορές πιστώσεων προς την Καταλωνία από την Ισπανική Κεντρική Κυβέρνηση. Επειδή φυσικά η συλλογή φόρων γίνεται από την κεντρική κυβέρνηση. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει λάβει υπόψη την ε, δυνατότητα τα προγράμματα αυτά που αναφέρατε αν μπορούν να αγοράσουν και ομόλογα από περιφέρειες, από περιφερειακές κυβερνήσεις και όχι μονάχα κεντρικές κυβερνήσεις. Παραγματικά χάρη αυτά της Καταλωνίας τα ομόλογα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το σύστημα αυτό αγοράς ομολόγων είναι σε λειτουργία για κάποιους μήνες. Βλέπω ότι τώρα όλες οι χώρες βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Όλες οι χώρες σε διαφορετικό βαθμό. Φυσικά ταχύτητος και άμεσης επιτυχίας. Όλες οι χώρες οι οποίες έπρεπε να προχωρήσουν σε προσαρμογές έχουν πάρει την απαραίτητη δράση και είναι όλες δεσμευμένες να προχωρήσουν και να αποδώσουν καρπούς οι προσπαθίες τους. Αυτό για το πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας. και τώρα θέλω να είμαι ίσως όχι αισιόδοξο γιατί αυτό θα ήταν υπερβολικό, αλλά τουλάχιστον να δείξω μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Αν δούμε ποια είναι η κατάσταση των δεσμεύσεων των χωρών μελών της ζώνης του ευρώ για να επανέλθει η σταθερότητα στον προϋπολογισμό τους, έναντι αυτού που κάνανε πριν από ένα χρόνο, θα έλεγα ότι είναι σημαντικές οι πρόσθετες προσπάθειες που έχουν γίνει. Για το δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας, Πρέπει να θυμόσαστε ότι το σύστημα αυτό για, τα, για τη σταθερότητα είχε σαν στόχο να εξασφαλίσει τη σωστή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής όταν υπήρχαν προβλήματα στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα στην οικονομία. Δεν είναι λοιπόν ένα σύστημα εξαγοράς ομολόγων της Α ή Β χώρας επειδή υπάρχει έλλειψη ρευστότητος εδώ ή εκεί αγοράζει ομόλογα το σύστημα αυτό όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική δεν λειτουργεί σωστά. Έχει παραλύσει, δεν μεταδίδεται σωστά, επομένως θα πρέπει να την επανααναζωογονήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. αυτό είναι ο κύριος λόγος ύπαρξης αυτού του συστήματος και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τον τελευταίο καιρό. Μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω τι σημαίνει την αναζωογόνηση των διάβλων νομισματικής πολιτικής. Αλλά, με λίγα λόγια, η αγορά κρατικών ομολόγων είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Είναι και ένας από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Αν αυτή η αγορά για μία χώρα, για δύο χώρες, για πολλές χώρες αρχίζει να έχει προβλήματα και να ε, να υπάρχει εμπλοκή και δεν μπορεί να λειτουργήσει ο μηχανισμός ε, νομισματικής πολιτικής. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το S&P. Δεν έχει άλλους στόχους. Η Ευχαριστώ Πρόεδρε Ντράγκη. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, Πρέπει να είμαι πιο δημιουργική τώρα στην ερώτηση μου τη δεύτερη, γιατί ήδη με κάλυψαν τι ερωτήσει. σω είναι σκληρότερη γι' αυτό η ερώτησή μου. Και ζητώ συγγνώμη. σαν αφορά νομισματική σταθερότητα και μακροπρόθεσμε διαθωτικέ μεταρρυθμίσει, είπατε εσεί επανειλημμένο ότι και η ανάπτυξη και άρα τα ωφέλη που ακολουθούν είναι από τι σημαντικότερε συνιστώσει για την αποκατάσταση τη απιστοσύνη των επενδυτών στην Ευρωζώνη. Και η ανάπτυξη είναι πολύ πιο εύκολη πάντα για μια χώρα όταν το νόμισμα τη είναι ασθενέστερο. Και ένα ασθενέστερο, με ασθενέστερη ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και ασθενέστερο ευρώ εναντί άλλων εξαγωγικών περιοχών ίσω θα βελτίωνε τι δυνατότητε ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Παρά τη μείωση ισοτιμία του ευρώ έναντι δολαρίου, είμαστε πάλι 8% πάνω το μέσο όρο από το 60 ευρώ ε, το 99. Άρα υπάρχουν ακόμα υπάρχει πίεση να μειωθεί η ισοτιμία. Είπατε βασικό στόχο είναι η σταθερότητα τιμών. Είναι εφικτό και ευκταίο να πετύχετε σταθερότητα στην Ευρωζώνη με, ε, ε, ε, με, χαμηλότερη ισοτιμία του ευρώ, τους, ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Απάντηση. Να πω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της και καλά. Είχαμε νομισματική πολιτική η οποία είναι ευέλικτη, υποστηρίζει τομείς που πρέπει, κυρίως την πραγματική οικονομία, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Είναι νομισματική πολιτική που ποτέ δεν λησμονεί. Έχει σαν πρωταρχική εντολή την εξασφάλιση σταθερότητας τιμών μεσοπρόθεσμα αλλά υποστηρίζει και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη. Τούτων λεχθέντων δεν έχουμε στόχους όσον αφορά την ισοτιμία, διότι αυτό δεν εμπίπτει εντός της βασικής μας εντολής που είναι να διατηρούμε μεσοπρόθεσμα τη σταθερότητα των τιμών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Πασκάλ ή Πασκάλ Ο Πασκάλ, συγγνώμη. Καλημέρα, καλησπέρα κυρία Πρόεδρε. Είπατε ότι αφορά την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και γι' αυτό δεν αγοράζει περισσότερα κρατικά ομόλογα. Θα λέγατε ότι η Αγγλική Τράπεζα και το Αμερικανικό Federal Reserve που έκανε το αντίθετο σήμερα δεν είναι αξιοπιστοί η θεσμοί. Δεύτερο στοιχείο αφορά τη Γαλλία. Πιθανότατα η Γαλλία θα χάσει το τριπλό α τις επόμενες ε, μέρες και εβδομάδες. Ποιες συνέπειες προβλέπετε όταν θα γίνει αυτή η υποβάθμιση με αρκετά ενδεχόμενα κατά ένα βαθμό, δύο βαθμούς, ε, μόνο η Γαλλία και άλλες χώρες. Λοιπόν, και το ερώτημα, εφόσον έχω 11 δευτερόλεπτα στη θέση μου. Μας είπατε επανειλημμένα ότι χρειάζονται εθνοτικέ ε, αλλαγέ για να βελτιωθεί η ανάπτυξη, να τονωθεί η ανάπτυξη. Μία από τι χώρε όπου οι εθνοτικέ μεταρρυθμίσει ήδη έλαβαν χώρα, η ΕΠΑ, διότι φαντάζομαι ότι τέτοιου είδους διαθωτικές αλλαγές έχετε υπόψη στην αγορά εργασίας. Έχει ΑΕΠ κατά κεφαλή που αυξήθηκε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως της Ευρωζώνης εδώ και 10 χρόνια. Ποια είναι η λογική διασύνδεση που σε επιτρέπει να πιστεύετε ότι οι εθνωτικέ μεταρρυθμίσει και απελευθέρωση αγορά εργασία επιτρέπει την ε, προώθηση τη ανάπτυξη, τη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Για το πρώτο ερώτημα η αξιοπιστία ενός θεσμού σαν την ΕΚΤ μετριέται με βάση τα αποτελέσματά της αλλά και την θεσμική της λειτουργία και πλαίσιο. Έχουμε μια εντολή που στοχεύει την σταθερότητα των τιμών. αλλά επίσης και μια εντολή που συνδέεται με την ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση. Άλλη είναι η εντολή του ΦΕΔ δηλαδή και άλλη η δική μας. Εμείς είμαστε περιορισμένοι στην αξι... στις τιμές, στη σταθερότητα των τιμών. Το ΦΕΔ συνδέεται μάλλον με την ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση. Άρα υπάρχει εδώ πολύ σημαντικός ρόλος του θεσμικού πλαισίου στο οποίο λειτουργεί το κάθε όργανο. Για τη Γαλλία, τι να σας πω. Δεν ξέρω αν η Γαλλία θα χάσει το τριπλό της α. Δεν θα το ευχόμουν, αλλά όπως είπα και πριν, δεν πρέπει να δίνουμε τόσο πολύ σημασία στις αλλαγές αυτές των αξιολογήσεων από τους οίκους. Και αυτό το λέω γενικότερα. Ούτε οι ρυθμιστές και επόπτες, ούτε ο οικονομικός τύπος δεν πρέπει να δίνουν τόση σημασία. Είναι απλώς ένα από τα δεδομένα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεν είναι τα πράγματα όπως πριν από 15 χρόνια, δεν είναι τόσο τρομερό. Αν χάσει το τριπλό της Α η Γαλλία, τότε θα αλλάξουν οι αξιολογήσεις και άλλων χωρών. Το θέμα είναι ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αν στο EFSF αν χάσει το τριπλό της Α η Γαλλία. Αυτό είναι το ερώτημα. Μπορούν να, μπορούμε να φανταστούμε διάφορα μέτρα αντιμετώπισης και τα επεξεργαζόμαστε εφόσον εμείς αυτή τη στιγμή λειτουργούμε το EFSF. Επεξεργαζόμαστε όλα τα πιθανά σενάρια, όχι μόνο της Γαλλίας. Βασικά όμως η δέσμευση του Συμβουλίου να λειτουργήσει πιο νωρίς το ESM από ό,τι προβλεπόταν. Και η ελπίδα, προσθέτω εγώ, στην ανακεφαλαιοποίησή του, η οποία και αυτή θα επιταχυνθεί, θα ήταν η σωστότερη δυνατή αντιμετώπιση σε οποιαδήποτε ζημία προς το EFSF θα προέκυπτε από τη μείωση της βαθμολογίας της Γαλλίας. Πρέπει δηλαδή να δούμε κατά πόσον το Μάρτιο θα φανεί αρκούν τα κεφάλαια του EFSF ή όχι. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Αυτό μπορώ να σας απαντήσω ως κοινά μέτρα προστασίας που μπορούμε να λάβουμε. Firewall. Δεν θα έλεγα όμως ότι είπα δεν χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι χρειάζονται. Αν αυτόν τον όρο τον εννοούμε μόνο ως μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, τότε συμφωνώ η αμερικανική αγορά εργασίας είναι πολύ ευέλικτη, ίσως και υπερβολικά για μερικούς. Γιατί πρέπει να δούμε πώς συνδυάζεται η ευελιξία με την αβεβαιότητα, αλλά στη ΗΠΑ όπως και στις άλλες χώρες χρειάζονται μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές. Δεν θέλω όμως εδώ να μιλήσω εκ μέρου του Ομπάμα και να του πω τι πρέπει να κάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο Μάρκος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώ ήλθατε στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σα ευχαριστώ που μιλήσατε και στα γερμανικά στην εισαγωγή σα. Αναφερθήκατε στο θέμα των εικόνων αξιολόγησης. Εγώ συμμερίζομαι την άποψή σας ότι δεν πρέπει να υπερτιμούμε αυτά τα οποία λένε οι οικοί αξιολόγησης. Αλλά χρειαζόμαστε και κάποιο γνώμονα, χρειαζόμαστε ένα μέτρο αξιολόγησης. Έχετε αποφασίσει για τρία χρόνια να δίνετε στις τράπεζες ρευστότητα με 1% επιτόκιο και επίσης μπορούν να καταθέτουν ως εγγύηση αξιο, αξιόγραφα τα οποία θεωρούνται δευτεροκλασσά, τα μικρότερης ε, φερεγγιότητος. Και επομένως αυτό είναι τμήμα της, ε, της ε, πρότασής σας. Αυτό όμως έχει νόημα να το κάνετε όταν δεν υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση για τους οίκους αξιολόγησης. Απάντηση. Καλό ερώτημα, διότι σαφώς πρέπει να πω ότι χρησιμοποιούμε αυτή τη, χρησιμοποίησαμε αυτή τις βαθμολογίες κατά το παρελθόν σαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά δεν είναι η μόνη μας ε, πηγή. Έχουμε δικές μας εταιρικέ ε, μεθόδους, δικό μας πλαίσιο, που, πώς να το πω, είναι ένα πλαίσιο που διατρέχει το σύστημα που έχουν οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες αρκετά ανεπτυγμένο. Πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ δύο ειδών αυ... αυξήσεως ε, των εγγυήσεων και των σχετικών αποφάσεων πήραμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε απόφαση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένα είδος εγγυήσεως από τριπλό α γίνεται δεκτό μέχρι να είναι απλό α. Αυτή είναι μια απόφαση και θα χρησιμοποιήσουμε τη δική μας αξιολόγηση. Σε τιμή αγορά υπολογίζουμε την εγγύηση και μετά εφαρμόζουμε κούρεμα. Η αξιολόγηση που κάνουμε είναι πολύ ε, συνετή, πολύ προσεκτική. Ε, υπάρχει μια άλλη απόφαση που πήραμε στον αφανάξη των εγγύσεων που κατά κάποιο τρόπο είναι καινοτόμα απόφαση. οι τράπεζες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις, τα δικά τους δάνεια προς, τις, προς τους πελάτες σαν εγγύηση. Αυτό απαιτεί να έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά κυρίως οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Γιατί Εθνικές. Διότι πολλοί ε, ε, έχουν καλύτερε γνώσει όσον αφορά τι επαφέ με του πελάτε. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν καλύτερε γνώσει. Θα ζητήσουμε λοιπόν από τι εθνικέ κεντρικέ τράπεζε τη δυνατότητα να αξιολογούν πιστώσει που δεν έχουν καν αξιολογηθεί από ε, οίκου αξιολόγηση. Υπάρχουν κάποιες λίγες ε, εθνικές κεντρικές τράπεζες που είχαν ένα τέτοιο σύστημα εσωτερικό αξιολόγηση για χρόνια τόσο πολύ που οι τράπεζες χρησιμοποιούσαν ε, τα δάνεια κατά το παρελθόν. Με διαφορετικό τρόπο, αλλά είχαν ένα παρεφερές σύστημα. Σε πολλές εθνικές κεντρικές τράπεζες αυτό το σύστημα δεν υπάρχει ακόμα. Άρα θα πρέπει να αναβαθμίσουν κατά κάποιο τρόπο τις υποδομές τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα. Εν τω μεταξύ, όλοι οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη διεύρυνση ε, επιλογών εγγυήσεων ε, θα, τον, θα είναι κάτι που θα αναλάβουν οι, Ευρωπαϊ... οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. Mm. Άρα οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα έχουν κάποια πρωτοβουλία στα χέρια τους όσον αφορά αυτό το κομμάτι ε, της αυξήσεως των εγγύσεων. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εκδώσει κατευθυντήριες, κοινέ κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό διότι δεν θέλουμε να έχουμε ε, διαφορές και διευθέτηση για όλα αυτά και θέλουμε να προστατεύσουμε και το δικό μας ισολογισμό καθώς και τον ισολογισμό των εθνικών ε, κεντρικών τραπεζών. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για το ίδιο θέμα αλλά με μια διαφορετική οπτική γωνία από τον προλαλήσαντα. Είπατε στις προηγούμενες απαντήσεις σας ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποφύγουμε υπερβολική συρρήκνωση της ε, ε, πίστοσης που θα έχει αποτελέσματα και στην ανάπτυξη. Πώς, το ερώτημα είναι πώς θα το κάνουμε αυτό αν δεν έχουμε σαφείς κανόνες για το πώς τα χρήματα τα οποία παίρνουν οι τράπεζες από τις τριετίες αυτές που λέτε πράξεις αναχρηματοδότησης με επιτόκιο μόνο 1% πώς θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά, μα δεν ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιούν οι τράπεζες, πώς θα ξέρουμε ότι αποφεύγουμε την, ε, το στέγνομα της πίστοση, αν δεν εξασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες χρηματοδοτούν πραγματικά την πραγματική οικονομία, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, που όπως είπατε προηγουμένω, πλήττονται από την έλλειψη ρευστότητα. Και τέλο, κύριε Πρόεδρε, πώ μπορούμε να εγγυηθούμε στον Ευρωπαίο πολίτη ότι στην Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο με το πρόγραμμα TARP, το Trouble Assets ε, ε, πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που δόθηκε για την αναχρηματοδότηση των αγορών πήγε σε μπόνους των υψηλών στελεχών. Και κάτι ακόμα, είπατε ότι η συρρήκνωση στις χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα θα πρέπει να είναι σύντομου χρονικού διαστήματος για να αποφύγουμε την πιστοτική συρρήκνωση, αλλά σε ορισμένες από αυτές τις χώρες και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, πέραν της εδραίωσης του προϋπολογισμού, υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα από την έλλειψη ρευστότητας που οδηγεί σε πολύ βαθύτερη ύφεση από ό,τι θα μπορούσε κανείς να προσδοκά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για το πρώτο σας ερώτημα. Είναι πολύ καλό το ερώτημά σας αν θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες που να διέπουν την λειτουργία των τραπεζών. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε κανόνες να λέμε στις τράπεζες τι ποσοστό θα πρέπει να επενδύσουν σε κάθε τομέα δραστηριότητάς τους. Στο παρελθόν, οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να αποφασίζουν τι δανείζουν στην πραγματική οικονομία, τι χρησιμοποιούν για λόγους χρηματοδότησης χάρη ε, αγορές κρατικών ομολόγων κτλ. Όλα αυτά βασίζονται στους δικούς υπολογισμούς σε ό,τι αφορά τη στρατηγική τους για τη σχέση κινδύνου με κερδοφορία για το επιχειρηματικό τους μοντέλο και όλα αυτά. Εδώ η δική μας ιδέα με την απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι να μειώσουμε την πίεση ε, χρηματοδότησης από ποσοτική έποψη και μειώνεται το κόστος χρηματοδότησης και ιδίως δίνεται στις τράπεζες μια μεσοπρόθεσμη προοπτική για τη χρηματοδότησή τους. Δηλαδή τους δίνεται μια εξασφάλιση ότι τουλάχιστον για τρία χρόνια θα έχουν αυτή τη γραμμή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να μην ξεχνάμε ότι η μέση διάρκεια των τραπεζικών ομολόγων που θα πρέπει να ξεπληρωθούν του χρόνου είναι περίπου τρία χρόνια. Γι' αυτό έχουμε πλησιάσει σε αυτό το επίπεδο. και τα ομόλογα αυτά για τις αγορές, οι αγορές ομολόγων έχουν ουσιαστικά σταματήσει να λειτουργούν εδώ και πολλούς μήνες. Οι περισσότερες τράπεζες δεν μπορούν να ε, εκδώσουν ομόλογα τα οποία δεν είναι του υψηλότερου επίπεδου ε, ασφάλειας χωρίς εγγύησης. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να έχουμε κανόνες για το πώς θα λειτουργούν οι τράπεζες σε κάθε χώρα θα πρέπει να είχαμε ένα πάρα πολύ πολύπλοκο πλέγμα κανόνων και σε αυτό το χρονικό σημείο η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα αποφύγουμε, θα αποτρέψουμε μια ύφεση που να οφείλεται σε έλλειψη χρηματοδότησης από περιστολή της ε, ε δανειοδότησης από τέτοιου είδου πίεση. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε να αποφύγουμε αυτό που είναι στις ΗΠΑ. Ξέρετε ότι πολλά έχουν γίνει στην Ευρώπη. Τα τελευταία, το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε πολλή δραστηριότητα των ρυθμιστών, των εποπτών. Όλοι οι εθνικοί επόπτες έχουν εκδώσει εντολές και κανονισμούς σε ό,τι αφορά την αμοιβή των στελεχών στις ε, τράπεζες. Υπήρξε καταρχήν μια γενική κατευθυντήρια γραμμή που συμφωνήσανε οι ηγέτες των G20 πριν από δύο χρόνια και στη συνέχεια έγινε δεκτή αυτή η απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ενσωματωθεί σε μια οδηγία για τα θέματα αυτά. Συνολικά λοιπόν, σε σχέση με την εμπειρία που αποκομίσαμε όλοι από την ε, κρίση στις ΗΠΑ, ήταν καλό αυτό. Δεύτερον, γιατί υπάρχει ένας άλλος λόγος. Οι τράπεζες δεν έχουν μοναχά έλλειψη πόρων, έχουν και έλλειψη ιδίου κεφαλαίου. Κάτι το οποίο δεν θέλουν να κάνουν τώρα είναι να κατασπαταλήσουν τις λίγες ευκαιρίες που έχουν να αυξήσουν το ποσοστό ιδίου κεφαλαίου τους δίνοντας υπερβολικά πριμ στους ηγέτες, στους αστελέχη Έχει αλλάξει λοιπόν τελείως το κλίμα από την εποχή αυτής της αρνητικής εμπειρίας στις ΗΠΑ. Συγγνώμη, είχατε και ένα τρίτο ερώτημα. Το τελευταίο μου σχόλιο, το τελευταίο μου ερώτημα ήταν ότι τα προβλήματα της ρευστότητος είναι αυτά στα οποία οφείλεται η πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ύφεση σε χώρες όπως η Ελλάδα. Το ερώτημα μου είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα στις χώρες αυτές που χρειάζονται πάνω απ' όλα ρευστότητα για να μπορέσουν να ξανααναθερμάνουν την οικονομική τους δραστηριότητα. Ναι, Νομίζω ότι οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής που πήραμε την τελευταία φορά, την προηγούμενη εβδομάδα, αντιμετωπίζουν και αυτό το πρόβλημα. Αλλά σε πολλές χώρες, πολύ, ένα μεγάλο μέρος της παροχής ρευστότητα γίνεται μέσα από ένα σύστημα έκτακτης παροχής ε, ε, ρευστότητας, οπότε είναι διαφορετικό αυτό από τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Η Σόφη. Ευχαριστώ. Κύριε Ντράγκη, είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε εδώ για πρώτη φάση στην Επιτροπή μας. Ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα. Πάντα υπάρχει η τάση να βλέπει κανείς τη λιτότητα και την ανάγκη διαθετικών μεταρρυθμίσεων από μια πολιτισμική πτυχή βορρά-νότου ή πολιτική δεξιάς-αριστεράς οπτική γωνία. Αλλά υπάρχει και άλλη πτυχή των γενεών. Και πολύ δισταγμή για μεταρρύθμιση και για μέτρα λιτότητας σχετίζεται με γενιές που δεν θέλουν να χάσουν προνόμια και ρίχνουν το βάρος σε νεότερους, σε μελλοντικές γενναίες. Το ερώτημά μου, πιστεύετε ότι γίνονται αρκετά, όχι μόνο από τις χώρες τις προβληματικές, αλλά ας πούμε και από τις καλές, ούτως υπήν, ε, σκανδιναβικές χώρες. Όσον αφορά συνταξιδότηση, μεταρρύθμιση στο συνταξιδοτικό τομέα, κάνουν αρκετά για να γίνουν βιώσιμα τα συνταξιδοτικά ταμεία μεσοπρόθεσμα. Και πιο συγκεκριμένα για τη χώρα μου, την Ολλανδία. Θεωρείται ότι το συλλογικό στεγαστικό χρέος που είναι το υψηλότερο στον κόσμο δημιουργεί έναν ιδιαίτερο κίνδυνο και πιστεύετε ότι αν οι πολιτικές που ενθαρρώνουν το ιδιωτικό χρέος δεν αλλάχθουν ότι η Ολλανδία θα έπρεπε να υποχρεωθεί να αλλάξει τους κανόνες και την νομοθεσία. Απάντηση. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, νομίζω ότι σχετίζεται περισσότερο με επανεξισορρόπηση των ανισορροπιών μεταξύ των γενεών. Δεν είναι, πώς να το πω, η γενική εικόνα στην Ευρωζώνη είναι υπέρ των παλαιών γενεών και οι νέες γενές έχουν τα προβλήματα. Δεν θέμα βαθμού. Σε κάποιες χώρες αυτή η ανισορροπία είναι πολύ μεγαλύτερη και βεβαίως αυτές οι χώρες τώρα δρούν, διότι πιέζονται. Από τις αγορές πιέζονται, από τις πολιτικές συνθήκες κλπ. Και κάνουν σοβαρά πράγματα. Είναι ευπρόσδεκτο όταν ακόμα και χώρες που δεν πιέζονται, κυρίως από τις αγορές, αναγνωρίσουν το πρόβλημα Δηλαδή, διάκριση κατά των νέων γενναιών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν έχω τώρα απάντηση διότι είναι ένα θέμα που φορά συγκεκριμένη χώρα, μπορώ να σας υποσχεθώ όμως κάτι, ότι απόλυτα εντάσσεται αυτό στο ESRB, δηλαδή ένα από τα θέματα που πρέπει να εξετάσουμε. Αφορά ενδεχόμενη συστημική ανισορροπία κάποιων χρηματοπιστωτικών διευθετήσεων σε κάποιες χώρες. Σας υπόσχομαι μια απάντηση όταν επανέλθω για να μιλήσω ε, υπό την άλλη μου ιδιότητα. Ευχαριστώ. Αλφρέντο Παλώνη. Ο Αλφρέντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δράση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα τελευταία δύο χρόνια ήταν επί δύο βασικών πτυχών. Από τη μία πλευρά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγόρασε περιορισμένε ποσότητε ομολόγων, κρατικών ομολόγων, δευτεροβαθμίων αγορών σε κάποιε χώρες Ευρωζώνη όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία. Δεύτερον, μείωσε το επιτόκιο. όλα αυτά ήταν χρήσιμα και εκτιμήθηκαν, δε Όμως, η σημερινή συζήτηση για την κρίση στην Ευρώπη μας δείχνει ότι το ευρωπαϊκό πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα πληθωρισμού πλέον, αλλά από ε, και έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης. Το ερώτημα που έχω κύριε Ντράγκη για σας. Ποιε άλλε πολιτικέ νομισματικέ θα μπορούσε να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να συμβάλλει στο να αντιστρέψει την παρούσα τάση του αποπληθωρισμού και τη ύφεση, με περαιτέρω μείωση των επιτοκίων και με χρηματοδότηση περιορισμένη του, τραπεζικού συστήματος για να αποφευθεί το μπλοκάρισμα των πιστώσεων για την πραγματική οικονομία, αυτά αρκούν για την παρούσα κατάσταση. Ή, και είναι ένα ερώτημα, κινδυνεύουμε να είμαστε αναποτελεσματικοί λόγω του προβλήματος της αναχρηματοδοτήσεως των τραπεζών. Και σήμερα είδα και στη δική σας συνέντευξη ε, ότι είπατε ότι ίσως να έχουμε καταλήξει μια κατάσταση σε μια προσέγγιση που είναι κάπως ε, εσφαλμένη. Απάντηση, ευχαριστώ. Πάνω απ' όλα, η πιθανότητα του πληθωρισμού δεν είναι πολύ μεγάλη, ε, για την ώρα είναι αρκετά περιορισμένη. Πώς απαντούμε, πάντα λέμε ότι ποτέ δεν προδεσμευόμεθα άμα ρωτάμε, όταν μας ρωτάνε εάν θα μειώσουμε ή όχι τα επιτόκια. Λέμε ότι ποτέ δεν πρόδεσμευόμεθα. Όσον αφορά για τη χρηματοδότηση της οικονομίας, τα μέτρα πήραμε την περασμένη εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι όπως έλεγα, επεκτείνουν τη ρευστότητα σε τρία χρόνια και μπορούν οι ε, τράπεζε που δανείζονται με κάποια επιτόκια να το αναπροσαρμόζουν. Να, θεωρώ ότι από αυτή την άποψη Κάναμε πολλά, όμως σε πάση περιπτώσει εμείς θα δούμε λίγο πώς πηγαίνουν τα πράγματα, πώς εκτιλήσονται, τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, τι γίνεται συνολικά στην οικονομία και θα δούμε μετά τι θα κάνουμε. Όμως θεωρώ ότι αυτό που έγινε ήδη είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λενάρντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για αυτά που είπατε και για τους οίκους αξιολόγησης και ευχαριστώ και τα εισηγητέ για, για, την, για, το, για την πρόταση. Νομίζω ότι ακολουθείτε μια ε, ε, λογική πριν από τα stress test των Ευρω... της Ευρωπαϊκής Αρχής, European Banking Authority και της έγκρισης αυτής, είχαμε το European Financial ε, Stabilization Facility. Ε, και αυτό επηρέασε και τις τράπεζες που εκτίθενται περισσότερο στα κρατικά ομόλογα. Μετά έπρεπε να αντιμετωπιστεί η επανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Όμως το πρόβλημα είναι ότι τα πάντα πήγανε διαφορετικά από αυτό που προβλεπόταν. Δηλαδή, πέρα το να παρατηρούμε ότι απαιτείται τώρα καλύτερο συντονισμό με τι ευρωπαϊκέ αρχέ, τι εποπτικέ. Σα ρωτώ τώρα πώ θα προχωρήσουν να κάνει επανακεφαλοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών. Απομένει ένα στόχο άμεσο και πώ θα εφαρμοστεί αυτό. Και σε αυτό το πλαίσιο πιστεύετε ότι είναι ένα πρόβλημα το αίτημα από τις τράπεζες να δημιουργήσουν διατραπεζικά ταμεία που θα αντιστοιχούν στο 1% των εγγυημένων ε, ε καταθέσεων ε, και αυτή η εγγύηση προβλέπεται εκ των προτέρων και μετά. Όπως είπατε, απάντηση, η σειρά δεν ακολουθεί τη σωστή φυσική σειρά. Σήμερα η διαδικασία της επαρκεφαλοποίησης των τραπεζών έγινε κάτι πολύ πιο δύσκολο ή πιο δύσκολο ας πούμε. Ε, όχι μόνο από αυτό που προβλεπόταν όταν το όλο εγχείρημα αποφασίστηκε, διότι η κατάσταση σήμερα είναι πολύ διαφορετική από πριν, αλλά έγινε πιο δύσκολο και συγκρίση από πώς θα ήταν αν το FSF ε, ήταν λειτουργικό, ήταν λειτουργία. Δεν υπάρχει εναλλακτική ότι οι τράπεζες πρέπει να κάνουν ανακεφαλοποίηση. Βεβαίως υπάρχουν διάφοροι τρόποι και χρόνοι για να γίνει αυτό. αυτό που κανείς δεν μπορεί να ευχηθεί είναι ότι οι τράπεζες θα κάνουν ανακεφαλοποίηση που θα αυξήσει τα capital ratios μειώνοντας τα δάνεια. Γι' αυτό επιμένουμε στο ότι οι τράπεζες θα πρέπει να επανακεφαλοποιήσουν μη μειώνοντας τα δάνεια αλλά περισσότερο προσπαθώντας να αυξήσουν το κεφάλαιο ε, για προκαθορισμένο ποσό, κατά προκαθορισμένο ποσοστό. Κάτι άλλο σημαντικό που βγαίνει από την ανακοίνωση της EBA είναι ότι αναφέρεται μόνο ότι θα κάνει ε, κανονικές δοκιμές τεστ τον επόμενο χρόνο. Δεν θα επαναληφθεί το εγχείρημα που έγινε εκτάκτος που αξιολογούσε τα κρατικά ομόλογα ανεξάρτητα τραπεζών που βρισκόταν. Αυτό θα πρέπει να το δεχτούμε θετικά και οι τράπεζες θα μπορέσουν να κάνουν ανακεφαλοποίηση χωρίς να πρέπει απαραίτητα να έχουν τον εφιάλτη άλλης δοκιμασίας που κρατά 4, 5, 6, αυτό που κάναμε κατά παρελθόν. Όσον αφορά το διατραπεζικό ε, ταμείο, όπως και το ερώτημα που έκανε η κυρία Εντβέλντ, είναι κάτι στο οποίο υπόσχομαι να απαντήσω υπό την άλλη μου ιδιότητα, διότι για την ώρα δεν γνωρίζω την απάντηση. Σαν πρόεδρος του Συμβουλίου Αξιολόγησης του Κινδύνου. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Η... Κυρία Βόρτμαν Κόλ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ως μία από τις εισηγήτριες του Sixpack μαζί με τη Σιλβί Γκουλάρ και άλλους, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για να δω πώς θα προχωρήσουν τα θέματα αυτών των έξι νομοθετικών ρυθμίσεων. Ο προκάτοχός ο, προκάτοχός ο κύριος Τρίσε, ήταν πολύ ανοιχτός για νομοθεσία σε σχέση με τα θέματα αυτά και έπαιξε μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του Six Pack. Έχω μερικά ερωτήματα λοιπόν σε σχέση με την πρόταση για αυτή τη νέα συμφωνία η οποία διέρευσε προς, το, προς τα μέσα ανημέρωσης. Μιλήσατε για την ενίσχυση της διαδικασίας ε, ε, υπερβολικών ελλημάτων, να ενσωματωθεί σε πρωτογενές δίκαιο ο χρυσός κανόνας. Επίση ζητήσατε μεγαλύτερη οικονομική και δημοσιονομική ολοκλήρωση βάσει του Six Pack. Η πρόταση αυτή όπως έχει αυτή τη στιγμή διατυπωθεί κατά την άποψή σα είναι ένα ουσιαστικό και αποφασιστικό βήμα προς το, προς το εμπρός. Να σας δώσω τρία παραδείγματα που έχω αμφιβολίες. Πρώτα απ' όλα, ο ρόλος των κρατών μελών αναφέρεται πολύ καλά, αλλά ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Επιτρόπου για τον προεπολεσμό και φυσικά και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραμένουν ασαφείς ή δεν αναφέρονται καθόλου. Δεύτερον, μια νέα, ε, ένα νέο πρόγραμμα εταιρικής σχέσης οικονομικής και δημοσιονομικής για τα κάτι μέλη εφαρμόζεται για τα προγράμματα σταθερότητα των κρατών μελών, ενώ τα προγράμματα σταθερότητα και ανάπτυξη για τα κάτι μέλη, όπω αναφέρονται στο Six δεν αναφέρονται καθόλου σε αυτή τη συμφωνία και δεν είναι σαφέ αν αυτή η νέα, αυτό το νέο πρόγραμμα εταιρική σχέση θα υπόκειται στην ίδια διαδικασία εποπτεία όπω το Six Και τέλο, η συμφωνία Europlus που θα τύχει συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών. Εμεί βλέπουμε από τι αιτήσει εκθέσει ανάπτυξη ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος. Αλλά τα θέματα μακροοικονομικής εποπτείας και το θέμα της ειδική πλειοψηφία ανάσχεσης δεν αναφέρονται, ούτε αναφέρεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Είναι λοιπόν αυτή η πρότασή σας στο τελικό δημοσιονομικό συμβόλαιο που ελπίζετε να υπάρξει για την ε, δημοσιονομική και οικονομική ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όχι, η απάντηση είναι όχι, λέει ο κύριος Ντράγκη. Είναι απλώς ένα πρώτο βήμα. Είναι ένα πρώτο, πολύ πρώτο βήμα από πολλές απόψεις. Είναι ένα πρώτο βήμα γιατί έχουμε πολύ δρόμο να διατρέξουμε και έχουμε πολλές δυνατότητες να βελτιώσουμε τα πράγματα. Μπορούμε να βελτιώσουμε το ρόλο που μπορούν να έχουν τα διάφορα θεσμικά όργανα. Μπορούμε <clears throat> να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όλα αυτά που είναι πολύ σημαντικά στο six Μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα λοιπόν που έχουν αποφασιστεί. Αλλά το οικονομικό τμήμα, το γεγονός ότι το οικονομικό τμήμα του six δεν αντανακλάται στις τωρινέ αποφάσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει παραγκονιστεί. Και γιατί μπορεί να επανέλθουμε στο six γιατί έχουμε πολύ δρόμο να διατρέξουμε και επίσης διότι το... μπορεί να υπάρξει και μια χωριστή συμφωνία. Εγώ λοιπόν δεν νομίζω ότι η... το δημοσιονομικό συμβόλαιο πρέπει να περιλαμβάνει μονάχα τη λιτότητα αλλά πρέπει να έχει και μεγαλύτερη ανάπτυξη, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, δηλαδή τις ιδέες που διέπουν και το οικονομικό τμήμα του ΖΙΚΣΠΑΚ που πρέπει να αντανακλώνται σε μια νέα συμφωνία. Υπερβάμος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε σε κάποιον προκάτοχό μου, απαντώντας, ότι η εντολή της Τράπεζας της Αγγλίας δεν είναι, και της ΦΕΝΤΕΝ δεν είναι η ίδια με της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά κάτι μου έλεγε ο προκάτοχός Έλεγε πάντα ότι δεν αξίζει το θέμα να διερωτηθεί κανείς ποια είναι η εντολή, διότι με διαφορετικές εντολές τελικά όλες οι κεντρικές τράπεζες ακολουθούσαν παρόμοιες στρατηγικές ε, όσον αφορά την νομισματική πολιτική. Υπάρχει κάτι που άλλαξε όσον αφορά αυτό. Δεύτερο ερώτημα αφορά την εντολή που θα δώσετε στον εκπρόσωπό σας στην ομάδα εργασίας που θα ξεκινήσει εργασίες της αύριο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης ε, τα αποφάσισαν αυτό. Όσον αφορά τη θεσμοποίηση κατά κάποιο τρόπο να συμπεριληφθεί στη συνθήκη το σύμφωνο Europlus θεωρείται ότι είναι καλή στρατηγική για να βγει η Ευρωζώνη από την ύφεση την οποία αντιμετωπίζει. Στο ίδιο πνεύμα θεωρείται ότι είναι νομικός συνεκτικό να καθοριστούν οι εξαιρετικές περιστάσεις ενώ ο όρος εξαιρετικές περιστάσεις εμφανίζεται ήδη στην ίδια τη συνθήκη και κανείς δεν ήθελε να το χρησιμοποιήσει. Κάποιοι από εμά ζητούσαμε παρόλα αυτά να χρησιμοποιηθεί. Και αντιθέτως η έννοια των διεθνωτικών μεταρρυθμίσεων έχει εισαχθεί άνευ πολιτικής συζητήσεως το τι αποτελεί μια διεθνωτική μεταρρύθμιση. Τέλος, όσον αφορά τον, ε, ε, τον άλλο κανονισμό, προσέχει ο κ. Κάμερον στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Δεν τολμώ να σας ρωτήσω επί τι πιστεύετε για τη δημιουργία ενός ε, Ταμείου Αποζημίωσης για την Ευρωζώνη. Αν θέλετε να απαντήσετε, είμαστε ευτυχείς βεβαίω. Μπορώ να σας ξαναρωτήσω ποια ήταν η πρώτη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση ήταν η εξή. Ο κύριος Ζανκλόντ Τρισέ όταν βρισκόταν στη θέση σας μας έλεγε πάντοτε ότι η ΕΚΤ ακολουθεί ακριβώς την πολιτική που της επιβάλλει η εντολή της. Εσείς τώρα μας λέτε ότι χρειάστηκε να αλλάξετε νομισματική πολιτική σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί έχετε διαφορετική εντολή από των Αμερικανών. Τι άλλαξε μεταξύ τρισέ ε και ημών με ύψιλον. Πάντοτε τα εργαλεία που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν διαφορετικά. Ακόμη και όταν ο προκάτοχός μου έλεγε έχουμε την ίδια νομισματική πολιτική με τη ΣΥΠΑ, διαφορετικά ήταν τα εργαλεία ή ο προσανατολισμός της ε, νομισματικής πολιτικής ήταν ο ίδιος και είναι Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα που χρειάζεται κάποια διόρθωση σε πολλά τμήματά του και μια οικονομική κατάσταση που τουλάχιστον στην Ευρωζώνη λόγω της δυνατότητας μείωσης των δανειοδοτήσεων μπορεί να βλάψει την οικονομία. Το δεύτερο σας ερώτημα στο δεύτερο ερώτημα απαντώ ναι, είπατε τι έκανε η διάσκεψη ως νέο νομοθετικό πλαίσιο και αν έχει συνταγματική προτεραιότητα εκείνο. Ναι, αυτό ήταν όντως το μεγαλύτερο έργο της σύμβασης, διότι διασφαλίζει έναν έλεγχο εξάντε που δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του δευτερογενούς δικαίου που παράγουν τα κράτη. Και το τρίτο σημείο, ο καθορισμός ή ορισμός των εξαιρετικών περιστάσεων έδειξε απλώς ότι χρειάζονται ακόμη πολλά να γίνουν για να υπάρξει πραγματική συνέπεια μεταξύ όσων έχουν ήδη γίνει και των νέων μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Λέει λοιπόν απλώς ότι χρειάζεται παραπάνω μέτρα. Όχι μόνο το εξάμετρο, αλλά και άλλα. Είναι πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Για το ΙΤΑΒ τώρα. Αν μπορούσαμε να επιστρέψουμε στη συνεργασία προς όφελος όλης της Ένωσης, καλύτερα θα ήταν από το να αντιδρούμε χωριστά. Απ' την άλλη, οι χώρες της Ευρωζώνης έχουν δικά τους χωριστά προβλήματα, όντως. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λύση σε αυτή τη δυσκολία της συνεργασίας όλων, αλλά ταυτόχρονα της αναγνώρισης του γεγονότος ότι τα προβλήματα της Ευρωζώνης είναι ιδιαίτερα σε αυτήν. Δεν είναι απλό το πράγμα. Το είδαμε και στις 9 Δεκεμβρίου. Το. Ότμαρ. Κύριε Πρόεδρε. Μιλήσατε για μια τομή στις αποβάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η αγορά δεν το είδε ακριβώς έτσι. Φαίνεται να αμφιβάλλει ότι η πολιτική υλοποίηση των αποφάσεων αυτών θα ακολουθήσει. Ποια είναι η άποψή σας. Και επίσης τι γίνεται για τα μέτρα που έχει να έχουν να κάνουν με τη στρέβλωση, δυνητική στρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ πλουσίων μεταξύ και ε, μεταξύ ισχυρών και ασθενών τραπεζών και τι επίπτωση θα έχει επίσης η μείωση των επιτοκίων για την Ελλάδα. Yeah, the, um... you're right. Απάντηση, δίκιο έχετε. Η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, αναγνωρίστηκε λιγότερο από τις αγορές και από την κοινή γνώμη από ότι τις άξιζε. Και αυτό που προσπαθούσα να πω σήμερα και λέω έκτοτε είναι ότι είναι ένα σημαντικότερο βήμα από αυτό που θεωρήθηκε και εκτιμήθηκε αμέσω μετά τη διεξαγωγή τη Συνόδου Κορυφή. Πιθανότατα, όταν έχει κανεί τέτοιο αποτέλεσμα, πρέπει να διαρωτηθεί ποιε ήταν οι προσδοκίε και κατά πόσο οι προσδοκίε ήταν πραγματιστικέ. Και νομίζω ότι οι προσδοκίες από τη Σύνοδο Κορυφής σαν την ασημένια σφαίρα που θα έλυνε το πρόβλημα υπήρχε σαν προσδοκία και δεν ήταν ρεαλιστική από την αρχή. Όταν κρίνουμε την πρόοδο θα πρέπει να τη συγκρίνουμε με τις προηγούμενες συνόδους κορυφής και την πρώτερη εξέλιξη της πραγματικής κατάστασης. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι η Σύνοδος Κορυφής ήταν ένα βήμα πρόοδου. Για το άλλο, όσον αφορά τη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ υγιών και μη υγιών τραπεζών, δεν το έπιασα το ερώτημα, με συγχωρείτε. Υπάρχει ο φόβος για, το, για την απαραίτητη αύξηση κεφαλαίου σε ορισμένε τράπεζες. Οι τράπεζες οι οποίες έχουν ε, μακροχρόνια κονδύλια και έχουν ε, ακολουθήσει σωστή, αξι, ε, σωστή αποταμίευση και κεφαλαιοποίηση είναι σε διαφορετική θέση από τις φτωχότερες, από τις τράπεζες που δεν το έχουν κάνει αυτό. Αν θα αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί λέτε ότι θα είναι σε δυσχερέστερη θέση, σε διαφορετική θέση. Διότι υπάρχουν ανησυχίες όπως είπατε. Ότι δεν είναι ισότιμες οι συνθήκες στο τραπεζικό σύστημα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό. Οι φυστάμενοι κανόνες και οι οδηγίες, οι κανονισμοί και οδηγίες δεν κάνουν διάκριση μεταξύ τραπεζών. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ε, ισότιμες συνθήκες. Όμως πρέπει να δει κανεί το πώς εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα από τις εθνικές εποπτικές αρχές. Αυτό πρέπει να εξετάσουμε, να δούμε αν πράγματι είναι ισότιμοι όροι ή όχι. Ευχαριστώ. Καλώς. Δύο τελευταίοι ομιλητής. Χούμπνερ και Φέιο. Η Ντανούτα Χούμπ. πρώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, η διαχείριση των κρίσεων σε διασυνοριακό επίπεδο. Εν μία νυχτή δημιουργήσαμε ευρωπαϊκή εποπτεία. Πολύ γρήγορα λάβετε υπόψη τη συνήθη ταχύτητα λήψης αποφάσεων, αλλά κολλησιεργούμε ε, όσον αφορά το, το διασυνοριακό μηχανισμό για επίλυση κρίσεων. Ελπίζουμε ευρωπαϊκό μηχανισμό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμμετείχε στο προνομοθετικό στάδιο. Είχαμε έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και συζήτηση εδώ και ένα χρόνο. Σας προβληματίζει αυτό σήμερα το ότι ακόμα δεν έχουμε αυτό το θεσμικό πλαίσιο και πώς βλέπετε το μέλλον όσον αφορά το θέμα. Απάντηση. Πράγματι, θα έπρεπε να πω όμως ότι υπάρχει και ένα σχέδιο οδηγίας για τη δημιουργία ενός διαμεθοριακού συστήματος επίλυσης για τον τραπεζικό τομέα. Έχουν γίνει πολλά πράγματα, όχι κατά ανάγκη στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο για επιλύσεις τραπεζών και άλλων πιστοτικών ιδρυμάτων, resolution δηλαδή, σε διαμεθοριακό επίπεδο. Πέρα λοιπόν αυτό που κάνουν οι εθνικοί ρυθμιστές και επόπτες θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί <clears throat> οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό των διαμεθοριακών επιχειρήσεων. Θα πρέπει από τη μία πλευρά να επιτύχουμε αλλαγέ στην νομοθεσία που θα επιτρέψουν στους επόπτες ή οποιουσδήποτε είναι υπεύθυνοι για την ε, διαδικασία εκαθάρισης των, των ιδρυμάτων αυτών ένα κάποιο επίπεδο διακριτικής ευχέρειας και επίσης να υπάρχουν οι λεγόμενες εν ζωή διαθήκες από την πλευρά διαφορετικών πιστοτικών ιδρυμάτων που να καθορίζουν πώς θα γίνει η επίλυσή τους. Όλα αυτά έχουν γίνει λοιπόν και υπάρχει και ένα σχέδιο οδηγίας ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει όμως να παραγνωρίσουμε την πολυπλοκότητα αυτού του εγχείρηματο. Πρέπει να σας πω επίσης ότι υπάρχει και πολύ καλύτερη συνεργασία μεταξύ εθνικών εποπτών αυτή τη στιγμή για την παρακολούθηση των καταστάσεων που ανακύπτουν. Αλλά δεν είναι εύκολο αυτό το εγχείρημα, όπως έλεγα προηγουμένως, γιατί όταν αντιμετωπίζουμε σε διαχείριση, διαχείριση κρίσεων που ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου υπάρχει διαφορετική νομοθεσία περιπτωχεύσεως σε κάθε χώρα. Η πτωχευτική νομοθεσία έχει βαθιές ρίζες στη θεσμική και οικονομική ιστορία κάθε χώρας. Επομένως, μια περίπτωση που πρέπει να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός επίλυσης διαμεθοριακού χαρακτήρα, θα πρέπει να εξασφαλίσει και την συνεκτικότητα όλων αυτών των διαφορετικών πτωχευτικών συστημάτων. Έχετε διαφορετικά δικαστήρια που είναι αρμόδια και έχετε διαφορετική, διαφορετική εποπτική λειτουργία σε κάθε χώρα οι επόπτες αυτοί θα πρέπει να συμφωνήσουν για τον κατάλογο, για την αξιολόγηση των πιστωτών οι οποίοι θα πρέπει να αποσημειοποιηθούν στην περίπτωση μιας πτώχευσης. Έχετε λοιπόν σε συνολικό επίπεδο την ανάγκη να ξέρετε ότι μια τράπεζα που έχει διαμεθοριακό χαρακτήρα και κινδυνεύει να πτωχεύσει, να εξασφαλίσετε ότι οι πιστωτές αυτής της τράπεζας θα αντιμετωπιστούν με, με ισότιμο τρόπο σε, από διάφορα δικαστήρια που βρισκόνται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς αντιμετωπίζουμε ένα πιο απλό εγχείρημα γιατί τελικά θα έχουμε μία οδηγία η οποία είναι πολύ δύσκολο το έργο της να μπορέσει να εναρμονίσει την πτωχευτική νομοθεσία στα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ο Διόγκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε Ντράγκη, θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ, να σας ευχηθώ την καλύτερη επιτυχία, τη μεγαλύτερη επιτυχία για την εντολή σας που μόλις ξεκινάει. Και έχω ένα ερώτημα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σε μια συγκυρία όπου έχουμε τόσα προβλήματα για το ενιαίο νόμισμα, όπου περνάμε μια κρίση δημοσίου χρέους, θα ήθελα να ξέρω αν συμφωνείτε με την ιδέα των ευρωομολογών ή των λεγόμενων ε, stability bonds, όπως είπε ο πρόεδρος της Κομισιόν, και αν αυτό, όπως κάνει η Κομισιόν με μια πράσινη βίβλο, αν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί και να εφαρμοστεί. Ξέρω ότι είναι δύσκολο ερώτημα να απαντήσετε εν συντομία, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ικανότητά σας. Είναι πάρα πολύ σύντομη η απάντηση που θα σας δώσω. Τα ευρωομόλογα μπορεί να έχουν νόημα μέσα σε μια δημοσιονομική ένωση. Αν δεν έχετε μια δημοσιονομική ένωση όμως, πρέπει να θέσετε το εξής ερώτημα. Θα ήταν εφικτό ένα σύστημα όπου οι χώρες από κοινού εκδίδουν ε, ομόλογα και έχουν πλήρη αμοιβαία εγγύηση, ενώ συγχρόνως οι δαπάνες τους αποφασίζονται χωριστά η κάθε χώρα λοιπόν καθορίζει τις δαπάνες της χωρίς να υπάρχει κάποια κοινή συμφωνία. Υπάρχει αυτό το βασικό λοιπόν στοιχείο αυτής της διαδικασίας. Όσο περισσότερες χώρες παραδίνουν την εθνική τους κυριαρχία σε σχέση με τη δημοσιονομική τους πολιτική και θέλω να κάνω εδώ μια στάση και να κάνω μια διάκριση μεταξύ δημοσιονομικής στάσης και δημοσιονομικού περιεχομένου. Όσο περισσότερο τα κράτη δίδουν την κυριαρχία τους, παρετούνται τις, τις κυριαρχίες τους, τόσο πιο επιτυχημένη θα είναι οποιαδήποτε μορφή ευρωομολόγων. Όσο λιγότερο γίνεται αυτό, για λόγους οι οποίοι είναι πολιτικοί, ποικίλοι λόγοι, όλο και μικρότερο θα είναι το κέρδος από μία μορφή κεντρικών ευρωομολόγων. Γιατί αν κάθε χώρα έχει το δικό της φορολογικό σύστημα και τις δικές της ταπάνες. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για ένα κοινό σύστημα εξασφάλισης. Είναι πολύ δύσκολο η μία χώρα να εγγυάται για τα οικονομικά μιας άλλης χώρας χωρίς να υπάρξει δημοσιονομική εναρμόνιση. Υπάρχουν ενδιάμεσα συστήματα, ε, μερικές ε, εγγυήσεις και όλα αυτά. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα επιλογών. Λοιπόν, σας λέω ότι όσο πιο μεμονωμένες είναι οι πολιτικές των χωρών στο δημοσιονομικό τομέα, τόσο πιο ε, αποσπασματικές θα είναι οι πολιτικές εγγύησεων και τόσο μικρότερα θα είναι τα ωφέλη. Και θέλω εδώ να συμπληρώσω και το προηγούμενο, <clears throat> προηγούμενη απάντηση που έκανα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποστηρίζει τα σχέδια της Κομισιόν για την διαμεθοριακή επίλυση τραπεζών. Υποστηρίζουμε τα σχέδια της Κομισιόν και επίσης υποστηρίζουμε την εργαλειοθήκη και την ανάγκη να έχουμε ένα μηχανισμό εξάντε για την επίλυση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κάτι που δεν είπα προηγουμένως. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τράγκη. Έχουμε τελειώσει τον πρώτο μας διάλογο στα νομισματικά θέματα. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Προσβλέπουμε στην επόμενη <clears throat> συνάντησή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο άλλο θέμα. Θα τα ξαναπούμε το πρωί.